Uh, uh, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τρεις η ώρα, οπότε αρχίζουμε. Καλώς ήρθατε όλοι. Πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Προτείνω το σημείο 2 να αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση, όπως και το 19 για την ε, αντιπροσωπεία στην ε, Αφρική. Εάν δεν έχετε αντίρρηση δηλαδή, τροποποιείται έτσι η ημερήσια διάταξη. Συμφωνεί. Ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Και περνάμε τώρα στο σημείο 3. Ο ήθιστη, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Καλώς ορίζω λοιπόν και όσους μας παρακολουθούν στις οθόνες των υπολογιστών τους. Είτε στο Μπλιάνα, είτε στο Ταλίν, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε οπουδήποτε. Έτσι έχουμε διαφάνεια στη συνεδριάση μας και έχουμε και διερμηνία στη διάθεσή μας. Και για να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες διερμηνίας σας παρακαλώ να μιλάτε ξεκάθαρα και αργά ώστε να περνάει πιο εύκολα το μήνυμά σας. Σημείο 4 και 5. Πρόκειται για μια κοινή συζήτηση για μια άλλη εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Δημοκρατία της Σιγκαπούρης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας, τον David Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι στην σύστασή μου προτείνω τη σύμφωνη γνώμη. Και αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως για οικονομικούς και γεωστρατηγικούς, αλλά όχι μόνο. Και το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω εδώ και το ξέρουν και οι συνάδελφοι είναι ότι πρόκειται για μια παλιά συμφωνία. Η συμφωνία δηλαδή ελεύθερων συναλλαγών ε, υπήρχε ήδη από το 2012 και άρχισε να ισχύει το 2013. Οπότε οι φίλοι από τη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης αναγκάστηκαν να περιμένουν πολύ μέχρι τώρα. Πρόκειται για ένα κράτος πόλη όπως πολύ σημαντικό λιμάνι στην νοτιοανατολική Ασία και μόνη της η Σιγκαπούρη έχει περισσότερο εμπόριο με την υπόλοιπη περιοχή από ότι περίπου όλες οι χώρες μαζί. 10.000 εταιρείε έχουν γραφεία εκεί και πολλές επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους εκεί. Η συμφωνία αφαιρεί εκτός από έναν όλους τους δασμολογικούς φραγμούς τα κύρια όμως ωφέλη δεν είναι δοσμολογικά, υπάρχουν και μη δασμολογικά, όπως είναι οι ενωσιακές δοκιμές ασφάλειας για αυτοκίνητα και μέρη αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά προϊόντα, επίσης υπηρεσίες και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ακολουθεί η συμφωνία αυτή τους κανόνες GATT. Επίση, όσον αφορά τι δημόσιε συμβάσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε σύγκριση με τι δημόσιε συμβάσει με, με 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω. Επίσης, οι ονομασίε πρόληψη επίσης θα κατοχωρηθούν. Είναι η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγών για υπηρεσίες και για ποτά σε όλη την περιοχή. Πρόκειται επίσης για μια συμφωνία σταδιακή που ενσωματώνει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πέφτουν οι προδιαγραφές, κάθε άλλο. Η Σιγκαπούρη θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρεί το δικαίωμα της ρύθμισης και την διαχείριση της αλίας και των δασών εφαρμόζει τα δικά τη πρότυπα σε όλα τα αγαθά και τι υπηρεσίε που απολύτω στην Ευρώπη, διατηρεί όμω το δικαίωμα ρύθμιση, δηλαδή εφαρμογή ψηλότερων προτύπων για την προστασία τη εργασία και του περιβάλλοντο. Όσον αφορά τα εργασιακά, η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει ε, την γλώσσα που χρησιμοποιούν οι συμβάσει του Διεθνού Γραφείου εργασία δεν έχει επικυρώσει τις συμβάσει για τις διάκρισεις και την ε, ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Και παραμένει και μία ακόμα για την υποχρεωτική εργασία. Είχαμε επαφές με τους συναδέρφους από τη Σιγκαπούρ και είχαμε συζητήσει αν μπορούν να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για την επικύρωση ε, γενικά του συνόλου της σύμβασης ε, του ILO. Ακούσαμε διάφορες εξηγήσεις για τις εργασιακές τους πολιτικές. Ελπίζουμε πάντως η Σιγκαπούρη να μπορέσει γρήγορα να επικυρώσει και αυτές τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η ομάδα μου, όπως ξέρετε, ζήτησε ένα μηχανισμό κυρώσεων. Δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτήν την ε, συμφωνία. Όμως μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει μια θεώρηση, μια ρήτρα μάλλον αναθεώρησης ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Επίσης, η συμφωνία επίσης που συμπεριλήφθηκε ε, συνοδευτικά με αυτή την πρώτη αναφέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι οικονομικές αξίες είναι βέβαια σημαντικές, αλλά η γεωστρατηγική σημασία είναι εξίσου σημαντική. Η συμφωνία αυτή θα είναι η πρώτη ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σχετική χώρα. Οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται με την Ινδονησία και μπορεί να συνεχιστούν και με την ε, Μαλαισία και την ε, Ταϊλάνδη και ελπίζουμε να συμπεριληφθεί και το Βιετνάμ σύντομα. Στόχος μας είναι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών να γίνονται αναπεριοχή. Επιπλέον συμμετέχει στο TPP, στο Block 11, η Σιγκαπούρη. Οι εταίροι μας προχωρούν και εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους όσον αφορά το εμπόριο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση μας με την περιοχή γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε υπό το φως αυτού στηρίζω την σύναψη της συμφωνίας αυτής ελεύθερων συναλλαγών. Θέλω βέβαια να ακούσω την άποψη των συναδέρφων. χωριστά. Θα τα δούμε τα δύο. Ωραία, ευχαριστώ. Πρόεδρος, τώρα σκιώδης εισηγητές. Ε, ο κύριος Νίγκαλα αντικαθιστά τον συνάδελφο. Ευχαριστώ. Όντω αντικαθιστώ τον συνάδελφο. Δεν μου έχει δώσει όμως κανένα σημείωμα, τίποτα, για να τον αντικαταστήσω. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα. εκ μέρους του αλλά να σας πω τι νομίζω ότι θα έλεγε. Γνωρίζω ότι το ΕΛΚ στηρίζει τις δύο αυτές εμπορικές συμφωνίες που είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να ολοκληρωθεί αυτή η εμπορική συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Και το θέλαμε, είπε και ο συγγετής για ποιο λόγο καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Είναι τόσα χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και η διαδικασία. Οπότε έφτασε η ώρα να ολοκληρωθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία και το ΕΛΚ να ξέρετε ότι θα στηρίξει, θα υπερψηφίσει δηλαδή. Και εδώ και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. άρα ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε όλοι, Συνεργαστήκαμε στενά με τον, ε, με τον ε, καθηγητή αρμόδιο γιατί σειρά ετών. Και είναι η τελευταία θητεία που θα προλάβουμε να δούμε να υπογράφεται αυτή η συμφωνία ε, πριν φύγουμε εμείς. Δεν το πιστεύω κιόλα. Ότι ο Ιζάν Κλωτικού και οι άλλοι έχουν δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσει αυτό. Ασχέτως λοιπόν των σημειώσεών μου, η ομάδα μου στηρίζει πλήρω τη συμφωνία αυτή και ευχαριστώ τον εισηγητή για όλη τη δουλειά και τι καλέ διαπραγματεύσει που είχαμε και που φρόντισαν να συμμετέχουμε διαρκώ. Σε πολύ καλή συνέντευξη με όλε τι ομάδε, συζητήσαμε όλα τα θέματα και προσπαθήσαμε να πετύχουμε συνενέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Νομίζω, όπω είπε και ο εισηγητή, επειδή ο κόσμο ανησυχεί πού το πάνε οι Ηνωμένε Πολιτείε εμπορικά και έχουμε γίνει λίγο παθητικό επιθετικοί ω προ τι απειλέ και τον τρόπο που αντιδρούμε. Και είδαμε τι έγινε με τον Τραμπ και τη συμφωνία ναύτα. Σημαντικό είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αυτό να κυρωθεί ω το δυνατόν πιο γρήγορα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα στη δική σα την ομάδα, αλλά νομίζω ότι εάν ε, πάρουμε κάποιε διαβεβαιώσει από τη Σιγκαπούρη θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία και να περάσει μάλιστα με ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστούμε για τους Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, όπως ο προηγούμενος συνάδελφος. Δεν θα σας εκπλήξει, εάν σας πω ότι η ομάδα μου είναι υπέρ της επιτάχυνσης της σύναψης των ε, Συμφωνίων Ελεύθερων Συναλλαγών που έχουμε μπροστά μας, επιτάπητος. Και είναι πολύ καλό το νέο σε ό,τι αφορά την συμφωνία αυτή με τη Σιγκαπούρη και η Ιταλική κυβέρνηση είναι υπέρ. Δίνει πράσινο φως. Ξέρετε ότι στην Ιταλία έχουμε μία αντισυμβατική κυβέρνηση. Δεν της αρέσουν οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες και οι παρατάξεις αυτού του κοινοβουλίου. Αλλά έχουν καταλάβει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ότι είναι μια συμφωνία που θα έχει μόνο ωφέλη. Είναι win-win η συμφωνία. Θα μπορούμε να εξάγουμε πολλά προς την Σιγκαπούρη και την οικονομία της. από τις πλέον προηγμένες και εξευρωπαϊσμένες ασιατικέ οικονομίε στην Νοτιοανατολική Ασία. Και ω προ το κράτος δικαίου και ω προ την αξιοκρατία και τόσα πολλά άλλα πρότυπα που έχουν κοινά μαζί μα. Δεν είναι ακριβώ αυτό που θα μα άρεσε, ακριβώ αυτό που θα θέλαμε, αυτό που είπε ο κ. Βίνκλερ, ότι κάποιε συμβάσει ακόμα δεν έχουν υπογραφεί, αλλά εάν δεν μπορούμε να συνάψουμε συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, α το κλείσουμε το μαγαζί εδώ στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ τη ε, σύμφωνη γνώμη για την ε, συμφωνία αυτή ελεύθερων συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη και όποια άλλη μπορέσουμε να προωθήσουμε πριν το τέλο αυτή τη θητεία. Ευχαριστούμε. Για, για του Πρασίνου, ο κύριο Ζαντό. Όντω, όντως, καλύτερα να είναι κανεί οικονομολόγο τη Σιγκαπούρη παρά δημοσιογράφο. Διότι η Σιγκαπούρη είναι πρωταθλήτρια στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, αλλά όχι στην ελευθερία του τύπου. Κάτι θα πρέπει να σα ανησυχεί και αυτό. Η Σιγκαπούρη είναι στι τελευταίε χώρε ε, στον κατάλογο όσων προστατεύουν την ελευθερία του τύπου. Για του οικολόγου αυτό είναι ένα θέμα. Ήδη ω προ ε, τα δημοσιονομικά και την οικονομία. Δεν σας διαφεύγει ότι ένας μεγάλος αριθμός οικονομολόγων σήμερα ε, προβλέπουν οικονομικό κράχ ή οικονομική κρίση κατά πάσα πιθανότητα της ίδιας ε, κλίμακας με το 2008 ή και χειρότερη. Και αν η Ευρώπη ήδη δυσκολεύεται να ξεφύγει από τον απόεχο της οικονομικής κρίσης το 2008, δεν ξέρω τι θα σήμαινε μια νέα οικονομική κρίση, πολιτικός και οικονομικός. Βρίσκω ότι σε αυτό το νέο ε, θέμα, το ντοσχέ, ο τρόπος που η Σιγκαπούρη πέτυχε να περιορίσει τη δυνατότητα αυστηρή πλησίωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι κάτι ανησυχητικό για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Δεν θα σταθώ στο κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο συνάδελφο Βίλτερ είπε πόσο το κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι επικοινωνιακού περιεχομένου και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα των συμφωνιών, διότι δεν προβλέπει καν ε, κυρώσει και θεωρώ ότι επ' αυτού το Κοινοβούλιο πραγματικά έχει παραγωνιστεί τελείω ω προ την τοποθέτησή του για το θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εμεί θέλουμε το κεφάλαιο αυτό να λάβει την ίδια σημασία με τα υπόλοιπα. Ιδάλω είναι να συνεχίζουμε να φλερούμε μεταξύ μα για τη σημασία του κλίματο, τη βιοποικιλότητα, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και για όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ η Αν για την voorzitter. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, το εμπόριο με την Σιγκαπούρη ε, ξέρουμε έχει περάσει από πολλά στάδια, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για να προχωρήσουμε με τις οικονομικές υπηρεσίες που αναφέρονται και με την ε, εποπτική εξαίρεση αυτό που με απασχολεί εμένα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προστασίας σε περίπτωση κρίσης. Αν, ας πούμε, υπάρχει πρόβλημα με μια τράπεζα. Δεν περιλαμβάνουμε εδώ το ίδιο περιλαμβάνουμε για την συμφωνία ΣΕΤΑ. Οπότε συνδέεται αυτή η εποπτεία με δοκιμές, με τεστ ή όχι. Υπάρχουν εξαιρέσεις επίσης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις. Ενώ υπάρχουν και ξένοι παράγοντες οι οποίοι εργάζονται εκεί. Είναι αλήθεια? Σωστά το καταλαβαίνω. Για μας οι εξαιρέσεις αυτές είναι επικίνδυνες. Για μένα είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση θέλω να τονίσω ότι η ρύθμιση των κρατών μελών πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Θέλω να ξέρω αν υπάρξει κρίση στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, τι θα γίνει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις εμείς. Και επίση θέλω να ξέρω αν μπορούν σε περίπτωση κρίσης οι χώρε αυτέ να προβούν σε αναδιάρθρωση, αν θα υπάρχει αρμπιτράζ ή όχι και ποια είναι τα κριτήρια που ισχύουν. Τι γίνεται με το δημόσιο χρέος. Και γιατί δεν έχουμε εδώ τις ίδιες ε, προδιαγραφές και προβλέψεις όπως έχουμε για τη ΣΕΤΑ στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ. Δεν θα σας εκπλήξει η κριτική μου απέναντι στη συμφωνία αυτή για τη Σιγκαπούρη και σας εθαρρύνω να διαβάσετε την έκθεση της Oxfam που λέει από τη Σιγκαπούρη στην Ελβετία η χειρότερη φορολογική παράδοση. Αν λοιπόν σήμερα ε, διαπιστώνουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επαναστατούν, αυτό γιατί συμβαίνει. Σημαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό γιατί οι πολυεθνικές δεν πληρώνουν φόρους. Αν υπάρχει λοιπόν μία εμπορική συμφωνία με έναν από αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους, καταλαβαίνετε ότι σήμερα το μήνυμα αυτό το πολιτικό που στέλνουμε στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ άσχημο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αντιταθούμε στη συμφωνία αυτή. Ξέρω ότι είναι μια συμφωνία που από το 2010 διαπραγματευόμαστε και τα περισσότερα επιχειρήματα που ακούμε σήμερα είναι ναι, αλλά υπάρχει ο Τραμπ. Ναι, το 10 όμως δεν υπήρχε ο Τραμπ. Και τώρα χρησιμοποιούμε τη μαριονέτα του Τραμπ ε, για να ορμήξουμε και να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερε εμπορικέ συμφωνίε. Μα δεν ήταν σε αυτή τη θέση ο Τραμπ, δεν υπήρχε τότε. Και όμω χρησιμοποιούμε τα ίδια επιχειρήματα όπω και τότε. Λοιπόν, το μήνυμα αυτό που περνάει στους Ευρωπαίους πολίτες είναι πολύ αρνητικό. Και επανέρχομαι και επί της ουσίας αυτό που είπε ο συνάδελφος Ζαντό για την ε, χρηματοπιστωτική ελευθέρωση. Αυτό είναι το πιο προβληματικό κεφάλαιο πηγαίνουμε προς μια απορρίθμιση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ενώ θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την αντίθετη πορεία. Έχουμε επίση ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωραία, θα μου πείτε, λέω πάντα τα ίδια και τα ίδια. Ναι, αλλά έτσι έχω μάθει εδώ ότι για να μάθει κανεί ε, χρειάζεται επανάληψη. Λοιπόν, έχουμε επαναλάβει ξανά ξανά και σε άλλη περίπτωση κερδίσαμε. Λοιπόν, τώρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για αυτό το κεφάλαιο, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά, ίσως κάποια μέρα καταφέρουμε να κερδίσουμε, να έχουμε εμπορικές συμφωνίες με κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη που να προστατεύουν όπως προσφέρεται προστασία και σε άλλα κεφάλαια. Στις επενδύσεις έχουμε προστασία ενώ για το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη δεν προχωράμε στο θέμα της προστασίας. Θα ήθελα λοιπόν να δίνουμε την ίδια σημασία στον πλανήτη, στα κοινωνικά δικαιώματα, όπως δίνουμε και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η κυρία Καλτον Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τα επιχειρήματα των τέρων μας από την Σιγκαπούρη, διότι τα τελευταία χρόνια εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έχουμε υποβάλει κάποιες προτάσεις σε μια συμφωνία, συμφώνησαν, το αλλάξαμε, επανήλθαμε με άλλες προτάσεις, το δέχτηκαν και αυτό έγινε πάνω από δύο ή τρεις φορές. Κάθε φορά υποβάλλουμε μια νέα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με αλλαγές και εκείνοι προσαρμόζονται και το δέχονται. Καταλαβαίνω λοιπόν και έχω κατανόηση για όλα αυτά τα επιχειρήματα που ακούω σήμερα, αλλά πραγματικά το πρόβλημα είναι ότι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αποφασίσει ποιοι είναι οι κανόνες στους οποίους θέλουμε να βασιστούμε. Δεν έχουμε βάλει τάξη στο δικό μας σπίτι. Και αυτό που είναι λυπηρό σε αυτή την ε, υπόθεση είναι από το 2010 δεν υπάρχει καμία απτή ε, βελτίωση όσον αφορά τις συμβάσεις και τα κοινωνικά δικαιώματα βάσει των προδιαγραφών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προτείνει το Διεθνές ε, Γραφείο Εργασίας. Αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά αυτά που ζητούμε, από το 2010 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απολύτως καμία κύρωση των τριών τελευταίων συμβάσεων. Είναι σημαντικές αυτές οι συμβάσεις, το δικαίωμα του συνεταιρίζεται, το δικαίωμα της μη καταναγκαστικής εργασίας. Πρόκειται για πάρα πολύ βασικά δικαιώματα στον τομέα της εργασίας. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό, όπως είπε και η Μαρή, ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε εξίσου τους επενδυτές, τους όρους ε, που προστατεύουν τους επενδυτές αλλά και τους εργαζόμενους, τους ε, πολίτες μας. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Παρόλα αυτά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ζητώ λοιπόν από όλους σας, αλλά και από τις αρχές της ε, Σιγκαπούρης, να στηρίξουν αυτήν την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Πιστεύω βεβαίως ότι θα πρέπει να δούμε μια κίνηση και μια πρόδροση όσον αφορά την κύρωση των συμβάσεων πριν υπογράψουμε εμείς την συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω και την υπογραφή αλλά και την εφαρμογή το συντομότερο δυνατό αυτής της συμφωνίας. Οι αρχές της Σιγκαπούρης περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι και από πέρσι που συνειδητοποίησαμε ότι η δυσαρέσκειά τους έφτασε μέχρι εμάς ε, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, έχουν δείξει μεγάλη υπομονή και κατανόηση και έχουν ε, προσαρμοστεί σε αυτά που τους ζητήσαμε πολλές φορές και πραγματικά η στάση τους είναι παραδειγματική. Έχουν ε, περιμένει ως, κάθε φορά που τους το ζητήσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και εμείς να κάνουμε μια κίνηση και να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Δεν πρέπει να περιμένουμε όλα να ικανοποιούνται ακριβώς όπως το έχουμε φανταστεί. Η Σιγκαπούρη, αν θέλετε, ήταν και ένας ουδέτερος χώρος, τον οποίο επέλεξαν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και οι δύο Κορέες για να συναντηθούν και να πλησιάσουν οι μεν τους δε. Πιστεύω λοιπόν ότι η Σιγκαπούρη έχει μία θέση στη διεθνή σκηνή. Υπάρχουν και άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνίες, οι οποίες δεν έχουν αυτή την ε, ίδια ε, τοποθέτηση. Και βεβαίως είναι διαφορετική χώρα από τις ευρωπαϊκές χώρες η Σιγκαπούρη, αλλά δεν μπορούμε να τους προσάψουμε αυτήν την διαφορά τους. Ε, θα πρέπει να είμαστε σαφείς, να υπογράψουμε και να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτήν τη συμφωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε θετικό πνεύμα και την ίδια ώρα να ακυρώσουμε βεβαίως την συμφωνία αυτή. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε με τη Σιγκαπούρη, καταλαβαίνετε ότι όλες οι υπόλοιπες ασχετικές χώρες θα περιμένουν πολύ παραπάνω. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να δείξει την αξιοπιστία και την ε, συνοχή στη στάση μας ε, στην περίπτωση αυτή. Εάν λοιπόν ε, θέλουμε την υπογραφή της Συμφωνίας της Εγκαπούρης, θα πρέπει να το συγκρίνουμε με αυτά που θυμήσαν οι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που παρενέβησαν. Δηλαδή ότι διαρκώς αλλάζαμε τα αιτήματά μας, ε, διπλωματευτήκαμε με έναν εταίρο που φάνηκε πρόθυμο να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα που διαρκώ αλλάζαμε. Είναι σημαντικό λοιπόν για την αξιοπιστία τη όλη μα ε, στάση να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Και επίση δεν μπορούμε να, παρα... να, ότι είμαστε σε ένα κόσμο απολύτως ε, απομονωμένο από όσα συμβαίνουν. δεν θα πρέπει να αποφεύγουμε τη σύναψη συμφωνιών. Ίσα ίσα σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε πόσο δυνατή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το Κοινοβούλιο, ε, ώστε να μπορεί να προωθήσει μια σειρά από δικέ του προτεραιότητε, προτεραιότητε εναλλακτικέ σε σχέση με όσα συμβαίνουν και ότι έχετε δυνατότητα να συνάπτει τέτοιου είδου συμφωνίε. Νομίζω λοιπόν ότι και από αυτή την προοπτική το γεωπολιτικό ε, πλαίσιο και σκηνικό δεν είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσαμε να του ε, διαχωρίσουμε από την αξιολόγηση, την πολιτική και την οικονομική της συμφωνίας που θέλουμε να εγκρίνουμε. μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο, ε, να δείξουμε ακόμα μεγαλύτερη πυγμή ε, στι στη με, τον εταίρο, με τους εταίρους μας από τη Σιγκαπούρη. Λόγω χάρη τα βήματα μπορούν να γίνουν για την κύρωση της σύμβασης του ILO, του Διεθνου Οργανισμού Εργασίας ή άλλα πρότυπα που αρχίζουν να γίνονται πρότυπα ε, σαφή. Αυτά είναι μια ευκαιρία να επιβάλλουμε τα πρότυπα αυτά και στις επόμενες φάσεις του διαλόγου με τους Σιγκαπουριανούς. Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία ως ένα ε, ε, βήμα, ένα εφαλτήριο για να υπάρξει συνέχεια στις προσπάθειες που γίνονται ε, με τη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε. Και η κυρία Μαρία Μάρτιν Πότα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συνοπτική. Καλωσορίζω την έκθεση του κυρίου Μάρτιν και τη σύσταση του το Κοινοβούλιο να δώσει συμφωνή γνώμη για τη σύναψη της συμφωνίας. Ξέρω ότι έχετε συζητήσει διαμακρών τα αίτια που θα έδειχναν ότι είναι καλή ιδέα να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και όπως είπε ο συγητής είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη όχι μόνο τους οικονομικούς λόγους αλλά και το γεωπολιτικό πλαίσιο. Και εδώ δεν θέλω να Ε, σταθώ ε, στην εχθρική στάση κάποιων από τους εμπορικούς μας εταίρους και να τους ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους. Απλώς είναι στιγμή τώρα να ε, προωθήσουμε τα πρότυπά μας, αυτά που θεωρούμε ορθά και να επιδιώξουμε την επιβολή του στην πράξη. Τη στιγμή που σε άλλες περιοχές του κόσμου αυτό το προσδοκούν από εμάς. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε λόγο στο ε, πώς θα πάνε τα πράγματα αυτά, τα διεθνή πράγματα. Είναι ευκαιρία. Η Σιγκαπούρη μας τη δίνει αυτή την ευκαιρία. Έχουμε εδώ την προληπτική στον προληπτικό διαχωρισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτι που θα επιτρέψει σε αυτό το σώμα να κοιτάξει κατά πόσον τηρούνται οι βασικέ γραμμέ τη σύμβαση του ΑΕΛΟ, αν υπάρχει συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και να μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στη Σιγκαπούρη. θα δούμε τώρα πώς ε, μπορεί να το προωθήσει αυτό η εισηγητής και να θυμίσω ξανά το ότι είναι σημαντικό να θέσουμε σε εφαρμογή τα πρότυπά μας και να συνάπτουμε συμφωνίες που τα εμπεριέχουν. Ίσως όλοι να επιδιώκουμε τον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικά μέσα. Πρόεδρος, ο κύριος Μάρτιν. Ναι, Νομίζω ότι βεβαίως και θα θέλαμε να κυρωθούν οι τρεις συμβάσεις ε, του ΑΕΛΟ από την ε, Σιγκαπούρη. Αλλά όχι μόνο. Εγώ πήγα στην ε, Σιγκαπούρη με αυτό κατά νου. Μίλησα και με τον Υπουργό Εμπορίου, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους το είπα με μεγάλη σαφήνεια. Και είχαμε κάποιες αιτιολογίες για ποιο λόγο δεν έχουν υπογράψει ακόμα. Παραδείγματος χάρη ε, όσον αφορά την καταργαστική εργασία. Και η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε εμά. Δεν λέω ότι ήταν ικανοποιητικέ, αν θέλετε, οι απαντήσεις. Ε, μιλήσαμε και για τους κρατούμενους και τα επιχειρήματα τα οποία μας ε, έδωσαν είναι ότι όλα αυτά δεν ε, αφορούν και δεν είναι το αντικείμενο της ε, σύμβασης ε, του ILO για την καταναγκαστική εργασία. Βεβαίως λοιπόν το θέμα των ωραρίων εργασίας, το θέμα της παρενόχλησης σεξουαλικής και άλλης, το θέμα των ε, κυρώσεων που επιβάλλονται και της ε, ποινικοποίηση κάποιων πράξεων ε, στις συμβάσεις εργασίας, το θέμα του περιορισμού σε κάθε είδους διαμαρτυρίας, απεργίας κτλ. Σίγουρα Πάντως από μέρους των αρχών της Σιγκαπούρης έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος και υπάρχει από τη μεριά τους βούληση να υπογραφούν οι τρεις αυτές συμφάσεις. Το 2017 στις 21 Ιουνίου η Σιγκαπούρη έχει υπογράψει την σύμβαση, την πολυμερή σύμβαση με τον ΟΣΑ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα φορολογίας. Και αυτό είναι κάτι που σαφώς βοηθάει για την πάταξη φαινομένων φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι για μια χώρα σαν τη Σιγκαπούρη με 5 εκατομμύρια κατοίκους, για μια χώρα που βεβαίως ε, δεν γνωρίζει την οικονομική κρίση που γνωρίζουμε εμείς και βεβαίως ε, το γεγονός ότι η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας ε, Ελεύθερου Εμπορίου από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο έχουμε καθυστερήσει από δικής μας πλευράς. Είναι κάτι που σίγουρα δεν έχει άμεση σχέση με την οικονομική κρίση. Πρόεδρος, προθεσμία για την ε, υποβολή των τροπολογιών είναι 9 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Και θα συνεχίσουμε με τις ε, προστασίες, με τα θέματα που αφορούν τη προστασία των ε, επενδυτών και Βεβαίως υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως ε, είπατε η Σιγκαπούρη έδειξε μεγάλη υπομονή στο θέμα της ε, συμφωνίας του ελεύθερου εμπορίου ότι φυσικά μετά την ε, αντικατάσταση του συστήματος ISES e από το ICS το 2014 έχουν ε, ενσωματωθεί όλα αυτά τα στοιχεία στο νέο σύστημα. Η Σιγκαπούρη σαφώς και είναι μία από τις χώρες με την οποία έχουμε μία ομαλή, αν θέλετε, κατάσταση όσον αφορά τις συναλλαγές και Βεβαίως το σύστημα ISDS και όλα τα άλλα συστήματα που σήμερα έχουν ενσωματωθεί και αντικατασταθεί από το IPA και το σύστημα ICS όπως έχει γίνει εξάλλου στη Συμφωνία ΣΥΤΑ και την σύσταση ενός ε, μικτού δικαιοδοτικού οργάνου το οποίο συνίσταται από δικαστές των δύο πλευρών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την προστασία των ε, δικαιωμάτων των επενδυτών και βεβαίως σε αυτή τις περιπτώσεις όπου δίνεται η δυνατότητα και στις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις να παρέμβουν, να υποβάλουν επιχειρήματα και στοιχεία και Υπάρχει και μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη ενός άρθρου για την ρύθμιση μέσω των ε, κυβερνήσεων του δημόσιου συμφέροντος, γιατί σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε να μην υπάρχει απολύτως καμία κυβερνητική και κρατική παρέμβαση. Η περίπτωση, αν θέλετε, στη Σιγκαπούρης, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι τόσο δύσκολη το σύστημα της ε, δικαιοσύνης στη χώρα αυτή λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός εμάς. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που έγινε και στην ε, Συμφωνία ΣΥΤΑ θα επαναληφθεί και εδώ για τους δικαστές, για να μην υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα και για τις περιπτώσεις δικαστών που έχουν αναλάβει περιπτώσεις που ε, παρεμβαίνουν ε, στις υποθέσεις και στις διαμάχες για θέματα και στις περιπτώσεις ε, της, των διαμαχών ISDS το σύστημα ICS και όπως έχουμε εκφράσει και στις άλλες περιπτώσεις παρόμοιων συμφωνιών, θα πρέπει σαφώς και να στηρίξουμε την συμπερίληψη όλων αυτών των στοιχείων. Βεβαίως και έχει σημαντική πρόοδο με τα νέα δεδομένα η συμφωνία αυτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα και βεβαίως η προστασία των επενδυτών, τα δικαιώματα των επενδυτών εδώ βρίσκεται στην καρδιά αυτού του θέματο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Κέλλη για δύο λεπτά. Πρέπει να πάω να ψηφίσω στην Ήτρε, λέει ο κύριος Κέλλη. Ο κύριος Καμάλ. Δεν λέω ότι θα είμαι πιο σύντομος από αυτό που μόλις είπε ο κύριος Κέλλη, αλλά πάσπερτος, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Λοιπόν, ελάχιστε διαφωνίε υπάρχουν ανάμεσα στην ομάδα μα και τον εισηγητή. Είμαστε ξεκάθαροι. Για άλλη μια φορά είναι το παλιό ζήτημα. Πώ συμπεριφερόμαστε στην Σιγκαπούρη, η οποία έκανε όλα όσα του ζητήσαμε. Του ζητήσαμε να ξανοίξουν ξανά και ξανά το θέμα και το έκαναν. Ωραία, υπάρχουν κάποιε διαφορέ για το ISDS. Καταλαβαίνω και την ερώτηση του εισηγητή που λέει Μα το χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά είναι μια ένα μοντέλο συμφωνίας προστασίας επενδύσεων που θα χρησιμεύσει και για άλλες περιπτώσεις. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι τη χρειαζόμαστε. Και ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία τους. Ο κύριος Τρουμός έφυγε. Τζάνικ. Α, ο κύριος Ζαντό, συγγνώμη, ο κύριος Ζαντό. Να ακούω σήμερα Βρετανούς, οι οποίοι αρνήθηκαν την κυδαιμονία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και προτιμάνε την διαιτησία των δικαστηρίων των πολυεθνικών, βρίσκω ότι πολιτικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, εγώ θα ήθελα να καταλάβω τι θέλουμε για βελτιώσεις στο σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτών κρατών. Μα εγώ φοβάμαι ότι κατά κάποιο τρόπο αν μου λέγατε ότι μπήκαμε στο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, εντάξει. Όμως, το ICS, το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, είναι ακριβώς το ίδιο με το ISDS. Είναι σαν να δίνουμε στις επιχειρήσεις και μόνο στις επιχειρήσεις ένα ειδικό καθεστώς σε σχέση με τις χώρες, σαν να τους δίνουμε προνόμια. Είναι κάτι απαράδεκτο δημοκρατικά. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε στους εκλογείς σας, στους συμπολίτε σας ότι εσείς δίνετε σε πολυεθνικές ένα τέτοιο καθεστώς και καταλαβαίνετε ότι ο κατάλογο των πολυεθνικών της Ζικαπούρης είναι τεράστιος. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση στον κόσμο που να μην έχει μια θηγατρική στη Ζικαπούρη. Οπότε εσείς αυτό που θα κάνετε είναι ότι θα δώσετε δικαιώματα σε πολυεθνικές που δεν δίνετε στα συνδικάτα, που δεν δίνετε στους καταναλωτές, που δεν δίνετε στους συμπολίτε σας. Στο σημερινό κόσμο λοιπόν ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να προχωράτε προς ένα τέτοιο σύστημα το οποίο δημοκρατικά είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο. Αν θέλουμε να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη των πολιτών αλλά η Ευρώπη των ε, επιχειρήσεων και των πολυεθνικών, πάρα πολύ ωραία. Αλλιώς όμως Πώ είναι δυνατόν να ψηφίσουμε μια τέτοια συμφωνία. Δεν έχουμε ακόμα εξάλλου την απόφαση του δικαστηρίου για την προσφυγή της Βαλονία αλλά και άλλων για το θέμα ακριβώς του κεφαλαίου για τις επενδύσεις. Οπότε, συγγνώμη, είναι παράλογο. Τι είναι αυτό το οποίο δικαιολογεί τον επιταχύνουμε την ψηφοφορία, ενώ από την άλλη περιμένουμε μια πολύ βασική απόφαση του δικαστηρίου για το ίδιο ακριβώ θέμα. Οπότε, συγγνώμη, εδώ πέρα αρνείστε διπλά τη δημοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι. Και στη σημερινή Ευρώπη, ειλικρινά, είναι κάτι απαράδεκτο πολιτικά. Ευχαριστούμε, Αν Μαρή Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κι εγώ θέλω να πω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να χειριστούμε αυτή την υπόθεση μέχρι να έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η συμφωνία με τη Σιγκαπούρη είναι η πρώτη ε, που συνάπτουμε βάσει των όσων προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνες. Ο Επίτροπος Ντεχούκ έχει εξηγήσει όλα αυτά και είχε πει ποιε είναι οι επιπτώσεις από τέτοιου είδου συμφωνίε. Το μέλλον του 2017 ακούσαμε ότι η προστασία των επενδύσεων είναι εθνική αρμοδιότητα. Παραμένει εθνική αρμοδιότητα και ότι κάθε τέτοια συμφωνία πρέπει να περνάει από τα εθνικά κοινοβούλια. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε, μάλλον γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, αποφάσισε και η Επιτροπή να βάλει το θέμα τη προστασία των επενδύσεων σε χωριστή συμφωνία. Το Σεπτέμβριο του 2017 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δέχτηκε μια προσφυγή από τη Βαλονία για το κατά πόσο στα πλαίσια της συμφωνίας ΣΕΤΑ όλα είναι σύμφωνα με τους κανόνες. Περιμένοντας αρνητική απάντηση. Μελετήθηκε το θέμα αυτό και υπήρξε και μια έκθεση η οποία κυκλοφόρησε. Η γνωμοδότηση πάντως αναμένεται ακόμα και φαίνεται ότι θα φτάσει του χρόνου η τελική απόφαση του δικαστηρίου, ίσως και μετά τις εκλογές. Αφορά ακριβώς το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων. Οπότε η Επιτροπή μας θα πρέπει να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου γιατί είναι κάτι πολύ βασικό όσον αφορά τα δικαιώματα θα πρέπει να περιμένουμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κίλτον Ντάρλινγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να θυμίσω ότι η μόνη φορά που ζητήσαμε από το ευρωπαϊκό κοινό την άποψή τους για την ατζέντα των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορηματικά απέρριψαν όσα πρότεινε ως προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έγιναν δημόσιας διαβουλεύσεις για το κεφάλαιο των επενδύσεων το τότε κείμενο της ΣΕΤΑ, ε, το κοινό ήταν απόλυτα αρνητικό, κατηγορηματικά μάλιστα. Ε, και σε σχέση με τα επιχειρήματα του Ντέιβιντ, θέλω να πω ότι για τη συμφωνία αυτή που θα αντικαταστήσει την τον τοξικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών με διμερείς συμφωνίες δεν μας ε, καθησυχάζει εάν κατ' επέκταση θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε ευνοϊκή πρόσβαση ε, στις πολυεθνικές για την επίλυση των διαφορών. Ε, πώς θα γίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει συμφωνήσει σε ένα κείμενο που έχει δεχτεί το όριμο και προηγμένο σύστημα, το δικαστικό σύστημα των δύο χωρών και παρόλα αυτά να επενδύονται, να, να προστατεύονται οι επενδυτές αλλά να μην υπόκεινται στο δικαστικό σύστημα των δύο εμπορικών εταίρων. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί ειδικό ευνοϊκό ε, για τις πολυεθνικές ε, εργαλείο και μηχανισμός με ολόκληρη γραφειοκρατία για να επιλύει αυτές τις διαφορές. Και τέλος, είναι κακή πολιτική λύση να γίνει δεκτή αυτή η συμφωνία. Είναι κακή πολιτική επιλογή, διότι δεν έχουμε ιδέα τι θα πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην αποφασή του για το κεφάλαιο των επενδύσεων, το ανάλογο τη ΣΕΤΑ. Ω πολιτικοί, άντρε και γυναίκε, το να υπερψηφίσουμε μια συμφωνία που μπορεί να ε, απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του χρόνου, είναι τελείω ε, επιζήμιο για την εικόνα μα. Ε, Α σκεφτούμε λοιπόν, άσχετα με το τι λέμε για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, δεν βλέπω κανένα λόγο να υποστηρίξουμε τη Συμφωνία για την Προστασία των Επενδυτών. Και πραγματικά ελπίζω ότι η πλειοψηφία στο ζώμα αυτό θα το απορρίψει κατηγορηματικά. Ευχαριστούμε ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να θα ήθελα να τα πω τα πράγματα και να είμαι λίγο πιο άνετος με αυτή τη συμφωνία, αλλά ανησυχώ. Ανησυχώ για να είμαι ειλικρινής και ο λόγος που ανησυχώ είναι γιατί Προσπαθούμε να προβλέψουμε ένα σύστημα επίλυση διαφορών για του επενδυτέ ε, δικαστικό ξεχωριστό. Είναι διαφορετικό αυτό από το αριστεία και έχω θέμα με το πώ ε, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με το θέμα αυτό. Ο λόγο που έχω πρόβλημα είναι ότι δεν θεωρώ ότι τα κράτη θα πρέπει να ορίζουν και να επιλέγουν δικαστές που μπορεί να έχουν ανάμειξη στις διαφορές. Ιδίω για κράτη που έχουν ε, δημοκρατικά διαπιστευτήρια. Νομίζω ότι είναι λυπηρό, αλλά και για τη Σιγκαπούρη ισχύει. Να αφήσουμε έξω από το δικαστικό σύστημα την πολιτική και τους πολιτικούς. Αυτός είναι ο στόχος. Και την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε για το σύστημα προστασίας των επενδυτών, νομίζω θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία, στα εδάφια του κειμένου που περιέχουν την ουσία. Τι είδου προστασία θέλουμε για τους επενδυτές. Καταλήγουμε να συζητάμε μόνο την επίλυση διαφορών και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ουσία του θέματο είναι μια συζήτηση που δεν την κάνουμε. Διότι αν δούμε τη βασική προστασία θα συμφωνούσαμε στο τι θέλουμε να προστατευτεί και τι όχι. Και αν δούμε αυτή τη βασική προστασία, τι είδου σύστημα διαιτησία ή επίλυση των διαφορών θέλουμε να δημιουργηθεί, νομίζω θα καταλήγαμε ότι το ICS είναι χειρότερη λύση από ό,τι ήταν το ISDS. Η δική μου μεγάλη ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πέσει σε μια ευρωπαϊκού τύπου παγίδα. Ένα πρόβλημα δική μα εσωτερική διαπάλυση με του σοσιαλιστέ δημοκράτε και το ανάγουμε σε πρόβλημα ευρωπαϊκή κλίμακα. Και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει το ευρωπαϊκό πρόβλημα παγκόσμιου ε, ε, βεληνικού. Ε, Λε και πρέπει να επιβληθεί αυτό το σύστημα σε όλο τον κόσμο. Ε, να μην ε, απορρίψουμε τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη μόνο για το ICS. Βέβαια, έχω και εγώ επικριτικά σχόλια, αλλά αυτό το σύστημα σίγουρα είναι ε, χειρότερο από τα SDS, αλλά καλύτερο από το τίποτα. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε σήμερα. Μαρία Ρενά. Ναι, όπως έλεγα και προηγουμένως, η επανάληψη βοηθάει στη μάθηση. Εδώ αναφερόμαστε πάλι στην προστασία των επενδυτών και θα ήταν ε, σωστό αν μπορούσαμε με ισορροπημένο τρόπο να προστατεύσουμε εξίσου και τα δικαιώματα των εργαζομένων και το περιβάλλον. Δεν θέλω λοιπόν κανένα σύστημα το οποίο δίνει πλεονέκτημα σε επενδυτές και μόνο. Η ερώτηση που υπευλήθη στο δικαστήριο από μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε την απάντηση του δικαστηρίου. Ίσως είναι λοιπόν λίγο νωρίς να ψηφίσουμε μία συμφωνία η οποία προβλέπει κάτι που δεν έχει αυτή τη στιγμή με σαφήνεια αποφασιστεί από το δικαστήριο. Περιμένουμε 10 χρόνια, όπως είπατε, πιστεύω ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Μπορούμε λοιπόν να δείξουμε ακόμα λίγη υπομονή, να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και να προσαρμοστούμε στην απόφαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Βίγκλα. Ευχαριστώ πολύ η επανάληψη, η επανάληψη και κερδίσαμε. Θα ακολουθήσω λοιπόν τη συμβουλή. Ο εισηγητής είπε πολύ σωστά νομίζω ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο ICS, το δικαστήριο δηλαδή που προστατεύει των επενδυτών καθώς και την ενίσχυση αυτού του συστήματος μέσω του δικαστηρίου αυτού. Νομίζω ότι και η Σκιώδης αλλά και ο εισηγητής το παρουσίασε σαν ένα ΣΥΤΑ πλάς. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή η κατάλληλη ώρα, αν θέλουμε να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας όλων αυτών των χρόνων, να ολοκληρώσουμε. Ναι, βεβαίως θέλουμε αυτήν την συμφωνία να εφαρμοστεί και αν υπάρξει, αν θέλετε, διάκριση των εξουσιών, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και το δικαστήριο θα κάνει τη δουλειά της και θα φτάσουμε στο τέλος ε, στα συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του δικαστηρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι ότι η Σιγκαπούρη έχει ή δεν έχει διμερείς συμφωνίες με κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα ICS θα ισχύσει είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη η Ρουμανία, είχαν τέτοιου είδου συμφωνίες πριν προσχωρήσουμε. Αυτές δεν εξαφωνίζονται από μόνες τους, αυτές θα πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτές οι παλαιότερες διμερείς συμφωνίες επενδύσεων με κάποιο τρόπο να σταματήσουν, δεν σταματούν από μόνες τους. Η κυρία Άουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που άκουσα. Ο συνάδελφος μίλησε κατά του ICS. Εν πάση περιπτώσει, η Σιγκαπούρη δεν νομίζω ότι ζήτησε αυτή την προστασία, αυτό το μηχανισμό προστασίας των επενδυτών, από ό,τι ξέρω. Είναι η 13η χώρα, από ό,τι ξέρω, όσον αφορά το κράτος δικαίου. Έχουν ένα σύστημα ε, δικαστικό το οποίο λειτουργεί με πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Γιατί λοιπόν θέλουμε αυτή την ε, συμφωνία. Συνάδελφοι, περιμένουμε το, την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι σωστό θα ήταν αυτή τη στιγμή να αναβάλουμε την δική μας απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ πολύ σύντομη θα είμαι. Από ό,τι φαίνεται, εδώ το θέμα της ισορροπίας και του κατά πόσο είναι δίκαιο αυτό το σύστημα για την προστασία των επενδυτών. Απασχολεί τους περισσότερους, ακούσαμε και τον εισηγητή και τον κύριο Βίγκλερ, που περιέγραψαν την κατάσταση και το ISDS είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και όπως ξέρετε η συμφωνία με την Σιγκαπούρη βασίζεται σε μία νέα προσέγγιση. Αυτό που θέλουμε σήμερα να αλλάξουμε είναι η νέα μας πολιτική να είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά τις επενδύσεις στο εξωτερικό. Και αυτή η συμφωνία με την Σιγκαπούρη ενσωματώνεται σε αυτήν τη νέα πολιτική. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα χρειαζόμαστε αυτήν την συμφωνία σαν ένα μήνυμα αν θέλετε ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των επενδύσεων. Αλλιώς επανερχόμαστε στην παλιά πολιτική όσον αφορά τις επενδύσεις. Για μας λοιπόν η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας με τη Σιγκαπούρη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα γιατί έτσι θα καταφέρουμε και με άλλες χώρες όπως το Μεξικό, το Βιετνάμ να δείξουμε ότι έχουμε μια νέα πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ισχύσουν αυτά τα νέα δεδομένα, αυτό το νέο δικαιοδοτικό όργανο, το πολυμερές και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρξει μια συγκεκριμένη συμφωνία με αυτήν την νέα πολιτική, αυτή τη νέα προσέγγιση. Και αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνει πολλά νέα δικαιώματα. Όσον αφορά την απόφαση που εκκρεμεί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Επιτρέψτε μου να σας ε, υπενθυμίσω ότι η Συμφωνία ΣΥΤΑ, την οποία έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εξηγήσουμε στις αρχές Σιγκαπούρης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει εγκρίνει τη Συμφωνία ΣΥΤΑ, εξαιτίας μιας εκρεμούς απόφασης που αφορά τη Συμφωνία ΣΥΤΑ δεν μπορεί να εγκρίνει τη Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης. Εδώ αναφερόμαστε σε μια συμφωνία η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί σε ισχύ πριν δοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, διότι όπως ξέρετε πρέπει όλα τα κρατημέλη να κυρώσουν την συμφωνία μέχρι να τεθεί σε ισχύ. Έχουμε λοιπόν το χρόνο, εάν η απόφαση του δικαστηρίου ε, μας υποχρεώσει να αλλάξουμε και να τροποποιήσουμε λίγο τα πράγματα πριν την εφαρμογή της. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ντέιβιτ. Για το τελευταίο, πρώτα απ' όλα. Για αυτά που λέει η Επιτροπή. Υπάρχει ένα επιχείρημα που θα ήταν να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά ώστε να μην εφαρμοστεί ακόμα η συμφωνία. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με τη συμφωνία ΣΥΤΑ το Κοινοβούλιο. Και θέλω να ενισχύσω αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να είχα πει και εισαγωγικά ότι σε αντίθεση με την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, εδώ χρειάζεται κύρωση από όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια, οπότε θα πάρει χρόνο. Έπειτα δεν υπάρχουν διαφωνίε σε εκκρεμότητα Μιλάμε για αυτό το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα πρέπει να περιμένουμε επίσης πολύ για να περιμένουμε το δικαστήριο. Τώρα, διάφοροι συνάδελφοι επανέλαβαν ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπήρχαν ήδη διμερείς συμφωνίες που ήταν ικανοποιητικέ. Έτσι έχει πει το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν και έτσι λέω και εγώ. Τώρα μπαίνουμε σε ένα νέο σύστημα. Και άκουσα τον Κρίστοφερ που είπε ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ήθελε την ε, συμφωνία τη ΣΕΤΑ, την είχαμε αρνηθεί. Για τη Σιγκαπούρα, συμφω... Σιγκαπούρη συμφωνώ με τους συναδέρφους ότι είναι γνωστή για το κράτος δικαίου. Είναι πάντα λεπτό και για μένα είναι πολύ εύκολο ε, να τα πω για την Επιτροπή, αλλά όπως είπα και πριν θα αποτελέσει μοντέλο αυτή η συμφωνία για μελλοντικές συμφωνίες με άλλες ασιατικές χώρες. Και η Σιγκαπούρη έχει καλό ρεκόρ ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν, κράτος δικαίου μάλλον, κράτος Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εμείς να λέμε αυτή η χώρα είναι εντάξει, άλλη δεν είναι. Τέλος, Εγώ δεν νομίζω ότι οι επενδυτές θα προχωρήσουν χωρίς να έχουν υποχρεώσεις και αυτοί από την πλευρά τους. Έχουν και εκείνοι όταν επενδύουν σε τρίτες χώρες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστούμε. Προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών είναι 12 Νοεμβρίου στις 6 το βράδυ. 12 Νοεμβρίου 6 μετά μεσημβρίας. Και έτσι ολοκληρώθηκαν και αυτά τα σημεία 6 και 7 και σε ένα λεπτό θα μπούμε στην ψηφοφορία. Ωραία. Είναι τέσσερις ακριβώς, οπότε αρχίζουμε τις ψηφοφορίες μας. Το πρώτο σημείο που θα ψηφίσουμε είναι το σημείο 8. Δασμολογικές ποσοστώσεις στον ΠΟΕ. Λόγω Brexit. Please. Έρχεται η κάρτα μου ηλεκτρονική, οπότε δεν μπορώ να συμμετάσχω στην ε, δοκιμαστική ψηφοφορία που θα κάνουμε, πάντω είναι στο δρόμο. Καλώ. Θα ελέγξουμε πρώτα τι κάρτες, πράγματι. Οπότε δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα απ' όλα. Ψηφίστε παρακαλώ. Everybody Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 31 παρόντες. Εντάξει. Οπότε, σημείο 8, κατανομή δεσμολογικών ποσοστώσεων περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε τις τροπολογίες της ΣΥΝΤΑ πρώτα απ' όλα. Εντάξει, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και μετά πάμε, άγκρι 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Άγκρι 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 4. Υπέρ, κατά, αποχές, ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για την 4, τροπολογία 4 Επιτροπής Γεωργίας. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Άγκρι 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα το σύνολο της ε, έκθεσης ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Μπράβο, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έχετε κάτι να ρωτήσετε. Να ρωτήσετε κάτι, εισηγήτρια. Εκτός μικροφώνου κάτι λέει, δεν την ακούμε. Νόμιζα ότι θέλατε να ζητήσετε την έναρξη των διαπραγματεύσεων, την εντολή. Ωραία, ναι. Η συγκήτρια όντω ζητάει εντολή για να αρχίζουν οι διοργανικέ διαπραγματεύσεις. Πρέπει και γι' αυτό να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Νομίζω ότι εντάξει, η συγκήτρια είναι υπέρ. Λέει ο πρόεδρος, τέλος της ψηφοφορίας με μεγάλη πλειοψηφία πραγματική για την εντολή αυτή. Ωραία, ευχαριστούμε. Και περνάμε στο σημείο 9, που είναι απόφαση για τη σύνεψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Συμβιβαστική αριθμός 5 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίθηκε. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 και 60 γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 62 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε για την 61. Καλώς. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Πράγματι. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 64. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 65. Α, 64 δεν φάνω πρώτος. 64. Ε, όχι, δεν την ψηφίζουμε. Ε, η 6 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ως προσθήκη η 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ως προσθήκη 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα καταπίπτει τη 96, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το ίδιο και με την 101. Ψηφίζουμε το δεύτερο της τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμφαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 113 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά.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 123 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και φτάνουμε στη συμβαστική 16 υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ως προστήκη ενδεχομένως 165 και 166 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνονται. Εκα... Απορρίφθηκαν, διορθώνω ο απορρίφθηκαν. 169 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 172 και 173 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ως προσθήκη 179 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 180. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 189 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα του 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2-2-6 υπέρ, κατά, από χέρ, απορρίπτεται. 2-2-7 υπέρ, κατά, από ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 2-2-7, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, εγκρίνεται. 2-2-8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ...231 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...μάλλον εγκρίνεται... ...αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά... ...αρχή της ψηφοφορίας... Τέλος. Εγκρίνεται. 2-3-2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2-3-3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Ελέγχουμε. 233 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος εγκρίνεται 2-3-4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2-3-5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε την 28 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 30. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνεται. Παρακαλώ πολύ, σηκώνετε τα χέρια σας. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται Το 44 δεύτερο τμήμα υπέρ. Μα, συγγνώμη, το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα του 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνουμε. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται τελική ψηφοφορία στο σύνολο του κειμένου πως έχει τροποποιηθεί αρχή της ψηφοφορίας τέλος 26 υπέρ ευχαριστούμε πολύ τον δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρόν στην ψηφοφορία διότι ακυρώθηκε η πτήση του. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Ξεκινάμε με την 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται επίσης. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 11 της ημερησίας διάταξης, το μέλλον της Ευρώπης. Πολύ σημαντικό θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται Οκτώ υπέρ κατά αποχές επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία Οκτώ υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ελέγχουμε την τροπολογία Οκτώ αρχή της ψηφοφορίας Τέλος. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 20 25 5, συμβαστική 5. Αποχές εγκρίνεται. 22, το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία σας παρακαλώ πολύ σηκώνετε τα χέρια σας Αρχή για την 27, αρχή της ψηφοφορίας, τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 δέλτα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 31 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε την 31. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Οκτώ συμβαστική υπέρ. Υπέρ της 8 κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές. Τι ψηφίζουν οι σοσιαλιστές. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την 37 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε αρχή της ψηφοφορίας για την 37 Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενδεκά συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Νομίζω ότι σώθηκε το μέλλον της Ευρώπης. Συγχαρητήρια. Okay, this concludes the voting session. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Θα διακόψουμε για ένα λεπτό. Όποιος θέλει να εγκαταλείψει την αίθουσα, παρακαλώ πολύ, με ησυχία. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η αποτίμηση της συμφωνίας για την ε, πρόσβαση της ε, Σαμόα στο εργαλείο προένταξης. Με συγχωρείτε συνάδελφοι, πάλι θα σας φάω τα αυτιά, αλλά όπως τα ξέρετε και εδώ πρότεινα την ε, σύμφωνη γνώμη μας για την πρόσβαση της ΣΑΜΟΑ ε, στο εργαλείο για την ε, προενταξιακή βοήθεια. Γιατί από το 2019 η ανεφδασμών, δεσμολόγητη ποσόσταση της Ευρωπαϊκής, της ΣΑΜΟΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αγορά της. Πρόεδρος, παρακαλώ σοπάστε. Και εγώ θα ήθελα να χαθώ το κύριο λέει ο κ. Από 1η Ιανουαρίου 2019 θα χάσει την αδασμολόγητη ποσοστοσή τη για προσβάση στην Ευρωπαϊκή Αγορά η ΣΑΜΟΑ, διότι υπάρχει το πρόγραμμα Τα πάντα εκτό από όπλα. Έτσι δεν θα υπάρξει διακοπή, εάν εγκρίνουμε το εργαλείο αυτό, στην, ε, εμπορικέ σχέσει τη ΣΑΜΟΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016 η ΣΑΜΟΑ επικαλέστηκε το άρθρο για τον αθλητικό εξοπλισμό και τον ε, εξοπλισμό ενόργανης γυμναστικής και ούτω καθεξής. Ο όγκος τέτοιων, εξαγωγών προς τη ΣΑΜΟ είναι πολύ μικρός. 5,5 εκατομμύρια ευρώ το 2017 για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της ΣΑΜΟΑς. Δεύτερος λόγος ήταν ότι υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για τις οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΑΜΟΑ με την ε, συμφωνία αυτή προενταξιακής βοήθειας. Καλύπτει μόνο εμπορικά αγαθά και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συμμετρικές απειλές της παγκοσμιοποίησης. Η ΣΑΜΟΑ έχει παγκοσμιοποιήσει το 86,8% των εξαγωγών της. Τα τελευταία 20 χρόνια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριο λόγο. Ε, φρέσκα λαχανικά και νοπά, αλκοολούχα και εινοπνευματόδη. 17,8% αποκλείεται όμως από, την, ε, ε από τις εξαγωγές. Είναι σημαντικά όλα αυτά λοιπόν για την ανάπτυξη της ΑΜΟΑ και την τοπική οικονομία. Υπάρχουν ε, σοβαρέ, σημαντικέ διατάξει για την προστασία του εμπορίου και βεβαίω οι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κάτω και τη δημοκρατία στοιχεία που τόσο άλλω επιβάλλονται λόγω τη συμφωνία τη Κοτονού. Και σε περίπτωση πρόληψη μέτρων, εάν παραβιαστούν όλα αυτά. Παρόλο που συμφωνώ ότι σε έναν τέλειο κόσμο αυτά δεν αρκούν, θα εκπνεύσουν όλα το 2020 και το ιδανικό θα ήταν, όπως συζητήσαμε με τον αυτή τη ΣΑΜΟΑ, είναι να λάβει μέτρα η ίδια η ΣΑΜΟΑ για πολλά θέματα όπως για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις κλιματικές αλλαγές με ευρύτερε μεταρρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή όμω αυτό δεν υπάρχει ως δυνατότητα γιατί τουλάχιστον συμμορφώνονται με την υπάρχουσα συμφωνία. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί με, το, με τα Φίτζη και τη Σαμόα τα θέματα και την Παππούα Νέα Γοηναία, ε, τα θέματα των κλιματικών αλλαγών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο ε, μεταξύ δεν βλέπω λόγο να μπλοκάρουμε την ευνοϊκή πρόσβαση της, Ευρωπαϊκ... της ΑΜΟΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πολύ αρνητικέ συνέπειε για μια τόσο μικρή οικονομία. Δεν βλέπω λόγο να μπλοκάρουμε τη συμφωνία και να έχουμε αντίθετη γνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και τώρα θα ψαρέψω τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής, ο κύριος Μάρτιν, ήδη ανέφερε ότι υπάρχουν ε, ανεπάρκειες στην ισχύουσα συμφωνία με τις νήσους του Ειρηνικού και θα πρέπει να έχουμε κάποιες δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διόρθωση των συμφωνιών και την κάλυψη των ανεπαρκειών. Να αναφέρω απλώ ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο εμπόριο και και βιώσιμη ανάπτυξη δεν υπάρχει κεφάλαιο για τις υπηρεσίε. Και μία σκέτη μνήμα στη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο αρχικό κείμενο που ανέφερε και ο Ντέιβιτ. Θέλω όμως να πω ότι από τις 5 Δεκεμβρίου 2017 η Σαμόα βρίσκεται στον αρνητικό κατάλογο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρα που δεν συνεργάζεται στα φορολογικά ζητήματα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει τι έχει κάνει εν ώψη τη συμφωνία αυτή. και με την ενδεχόμενη προσχώρηση της ΑΜΟΑΣ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Ρενά. Η κυρία Φορέντσα κάπου αναφέρεται ως κοιόδης, αλλά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την ενδιάμεση αυτή η συμφωνία εταιρική ε, σχέσης. Η Σαμό είναι μια πάρα πολύ μικρή χώρα, σαν το Λουξεμβούργο που είναι δικιά μας μικρότερη χώρα μέλος. Η Σαμό όμως είναι φορολογικός παράδεισος. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν με τη συμφωνία αυτή να διευκολυνθεί η μεταφορά παράνομου χρήματος. Οπότε πρέπει να δούμε η συμφωνία αυτή κάνει κάτι για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Έπειτα ο εισηγητής λέει ότι δεν υπάρχει ομάδα εσωτερική συμβούλων και δεν μιλάει καν για να δοθεί συνέχεια. Γιατί να μην υπάρχει μια προϋπόθεση προκειμένου να συνεχίσουμε με αυτή τη συμφωνία. Κλίμα, δικαιώματα ανθρώπων, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι πράγματα πολύ σημαντικά. Η ανάπτυξη αυτής της μικρής χώρας είναι βέβαια κάτι σημαντικό, αλλά σημαντικό είναι επίσης να καταπολεμήσουμε αυτά τα οποία παραβιάζουν τις αρχές μας. Εξού και δεν θα συμφωνήσουμε με αυτή την ε, συμφωνία μέχρι να υπάρξει νέα φορολογική ρύθμιση στη χώρα που να αποφεύγει αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ που τα προβλέπει αυτά. Οπότε νομίζω προς το συμφέρον όλων των πλευρών είναι να συμμορφωθεί η ΣΑΜΟΑ με καλύτερες προδιαγραφές. Τώρα είναι η Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, ο Ντέβιτ Μάρτινς ανέφερε τις εξαγωγές ε, μηχανημάτων γυμναστικής. Εγώ ρώτησα τον πρέσβη της ΑΜΟ που δεν καταλαβαίνει τα νούμερα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση και δεν βλέπει γιατί ο κλάδος αυτός πλήττεται από τη συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται μάλλον για μηχανήματα τα οποία πήγαν και ήρθαν από τη ΣΑΜΟ. Γι' αυτό θέλω περισσότερες επεξηγήσεις. Γι' αυτό. Δεύτερον, αν αφαιρέσουμε ε, τον κλάδο των μηχανημάτων αυτών γυμναστηρίου, μένουν οι πρώτες ύλε και η διατροφή. Άρα δεν υπάρχει διαφοροποίηση των εξαγωγών μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη. Οπότε αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης πώς θα βοηθούσε τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της ΑΜΟ προς την Ευρώπη. Απ' την άλλη βλέπουμε βέβαια το ενδιαφέρον που έχει η συμφωνία προκειμένου τα ευρωπαϊκά ε, προϊόντα να μπαίνουν χωρίς δασμούς στη Σαμόα. Όμως έτσι η φτωχή αυτή χώρα ε, θα έχει λιγότερα έσοδα. Πώς θα γίνει η αντιστάθμιση αν η χώρα αυτή δεν κάνει εξαγωγές προς εμάς. Ο ισολογισμός είναι έτσι αλλιώς ελληματικός ο εμπορικός. Οπότε στη συμφωνία αυτή δεν βλέπω αν υπάρχουν πράγματα τα οποία να ευνοούν τις εξαγωγές τους. Και τελειώνω με το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω ήθιστε χρησιμοποιεί ένα μέσο το οποίο είναι δασμολογικό. 1η Ιανουαρίου δηλαδή η Σαμόα δεν θα έχει πια προτιμησιακούς δασμούς προς την Ευρώπη, οπότε χρησιμοποιείται αυτή η πίεση ώστε η Σαμόα να ανοίξει τις πόρτες της χωρίς όμως να υπάρχει αντιστάθμισμα. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια σχέση από την οποία όλοι έχουν να κερδίσουν για μια χώρα τόσο ευάλωτη, ενώ η Ευρώπη είναι πολύ πιο δυνατή δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι μια δίκαια και καλή σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Ευχαριστούμε. Με κυρία Ζαρμέ τώρα. Ευχαριστώ κι εγώ. Πέρα από όλε αυτές τις σκέψεις και συμφωνώ απόλυτα, η Σαμόα είναι στο μαύρο κατάλογο των φορολογικών παραδείσων που έχει κονίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως μην ξεχνάμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία δεν γίνονται σεβαστά εκεί. Και μετά από μία έκθεση ε, τη Γερουσία, είδα ότι δεν ε, επηρεάζεται καθόλου η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα παιδιά από ό,τι φαίνεται δεν προστατεύονται παρκώς από τη βία, κάθε μορφή, είτε πρόκειται για σεξουαλική δηλαδή ε, όκληση ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι προχωράμε με δύο ταχύτητες. Και εσείς από ό,τι φαίνεται κλείνετε τα μάτια. Ιστορικά, γεωγραφικά, πράγματι, η ΣΟΑ μπορούμε να πούμε ότι οικονομικά είναι ένα παράρτημα της Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας, γεωγραφικά και ιστορικά. Και η Νέα Ζηλανδία που ήταν απικιακή δύναμη έχει πράγματι ιδιαίτερες σχέσεις με τη Σαμόα. Και έρχομαι στο δεύτερο ή το σπάδο προτελευταίο μου σημείο. Αυτή η συμφωνία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ε, μία πόρτα από την οποία θα μπουν διάφορα θα περάσουν διάφορα προϊόντα της Νέας Ζηλανδίας προς την Ευρώπη, χωρίς ποσοστώσεις. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι. Βλέπω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του 2018 στη δεύτερη σελίδα και βλέπω ότι δεν υπάρχει ποσόστοση σε αυτή τη συμφωνία. Η Νέα Ζηλανδία δηλαδή και η Αυστραλία μέσω της ΑΜΟΑ μπορούν ε, κάλλιστα να πλημμυρίσουν τη δικιά μας αγορά με προϊόντα τους. Δεν ξέρω, κλείνετε τα μάτια, προσπαθείτε να διακανονίσετε κάτι το οποίο όμως δημιουργεί ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και επανέρχομαι και στο αποτύπωμα άνθρικα. Σε αυτή την οικολογική μετάβαση που θέλουμε να κάνουμε. Σήμερα τελικά πουλάμε τις μεγάλες μας αρχές υπέρ της παγκοσμιοποίησης και του κέρδους. Το ξέρουμε, οι οικονομολόγοι, οι ειδικοί συμφωνούν σε αυτό, ότι η γη μπορεί να προσφέρει 2 με 3% των πόρων. Με τις συμφωνίες αυτές καταλήγουμε στο 116. 116 συμφωνίες έχουμε με τις οποίες, και τελειώνω, εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Σήμερα ζητάμε από τη γη να μας προσφέρει 12 με 13%. Χρειάζεται περισσότερη ταπεινοφροσύνη από τη δικιά μας την πλευρά και περισσότερη λογική. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Ερικα Σκόλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ Όλου και του εισηγητέ για την θετική, τον εισηγητή για τη θετική του αποτίμηση. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορικών Θεματών που είχαμε σε συνεργασία με εκπροσώπους από την περιοχή του Ειρηνικού, από την Παππούα Νέα Γουρινέα και το Φίτζι, στις 4 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη συνάντηση ε, τα νησιά της Αμόας και Τόγκα ε, που ενδιαφέρονται μόνο για αυτό το εργαλείο προνταξιακής στήριξη, είπαν μετά από συζήτηση ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστεί τέτοιο μηχανισμό. Μηχανισμό συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση τη υλοποίηση και του αντικτύπου αυτή τη συμφωνία. Και πραγματικά η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι εμπορικοί στόχοι και τη βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκονται με αυτή τη συμφωνία. Τα συμβαλόμενα μέρη επιμένουν στη δέσμευσή τους να εργαστούν για να προωθήσουν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τους στόχους της, δηλαδή τις βασικές εργασιακές συνθήκες και πρότυπα, το περιβάλλον, την σωστή διαχείριση των πόρων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ένωση ως Επιτροπή να υποβάλει γραπτή πρόταση για τη διαδικασία κοινή παρακολούθησης και την αξιολόγηση των ε, συμβαλωμένων μερών στην επόμενη συνεδρίαση Επιτροπής. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Ε, τα συμβαλώμενα μέρη σημειώνουν και την τοποθέτηση της Επιτροπής, της Επιτροπής ε, από το Κοινοβούλιο Θα φροντίσουμε οι μέρη σας να καταγραφούν ε, στο τελικό κείμενο της ε, συμφωνίας μαζί με τη ρήτρα για, τα, για την κοινωνία των πολιτών και μας ενδιαφέρει να παρακολουθείτε η συμμετοχή της κοινωνίας ε, των πολιτών όπως είπα και θα υπάρξει σχετική πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση. Ως προς τις συγκεκριμένες ζήτρες για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη τα συμβαλόμενα μέρη είναι περισσότερο ευνοϊκά στην ιδέα ότι πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση και να εξεταστούν τα πράγματα περισσότερο λεπτομεριακά. Μας ενδιαφέρει και τι γίνεται με τις συμφωνίες ε, μετά την Κοτονού, για τη φάση μετά την Κοτονού. Συμφωνίες που έχουμε αρχίσει να διαπραγματευόμαστε ω προ τι κοινέ του διατάξει και θα αρχίσουν να ισχύουν για όλε τι χώρε τη Καραϊβική και του Ειρηνικού. Ε, μαζί με τι συμφωνίε πενταξιακή βοήθεια. Θέλουμε να είναι αυστηρέ οι διατάξει για το εμπόριο, την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Και αυτή τη στιγμή οι συμφωνίε για τη φάση μετά την Κοτονού ε, προχωρήσει και εκπνεύσει, τότε θα χρειαστούμε να κάνουμε τεχνικές προσαρμογές σε αυτή τη συμφωνία. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και θα δούμε που βρισκόμαστε σε σχέση με τις διατάξεις αυτές. Σε ό,τι αφορά το θέμα φορολογικού παραδείσου και αρνητικού καταλόγου, είναι εκτός του πεδίου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, αλλά και στη συνάντηση που είχαμε με τους εκπροσώπους της ΑΜΟΑΣ, στο πλαίσιο της Επιτροπής για τη Συμφωνία. Δεσμευτήκαμε να συζητήσουμε το θέμα και η Σαμόα μας έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα αρχίσει να ασχολείται σοβαρά με το θέμα. και ότι εργάζεται επικοδομητικός προς την εξέβρεση λύσης. Αυτό το πενταξιακό εργαλείο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλου τομεί, όπω οι υπηρεσίε αργότερα, αν το ζητήσουν οι εταίροι. Άλλωστε, η Παππούα Νέα Γουινέα ήταν το πρώτο συμβαλόμενο μέρο σε τέτοια είδου συμφωνία ε, και έχει εκφράσει ενδιαφέρον στο να περάσει σε διαπραγματεύσει μαζί μα για το θέμα αυτό. Η πρώτη προτεραιότητα είναι τώρα η υλοποίηση τη υπάρχουσα συμφωνία και να δούμε τις ενταξιακές διαδικασίες και τις προενταξιακέ στη φάση μετά την Κοτονού και σε άλλους ενδεχομένω τομεί όπως οι υπηρεσίε. Σε ό,τι αφορά την διαφοροποίηση. Πολύ καλή παρατηρήσή σας και ευχαριστώ. Θα έλεγα ότι είναι πραγματικά εταιρική σχέση που έχει ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Η συμφωνία αυτή ήδη έχει βοηθήσει όσου έχουν συμπληθεί και την εφαρμόζουν σωστά, όπω η Παππούα και η Νέα Γουινέα, που είναι αφοσιωμένο, φανατικό εφαρμοστή τη συμφωνία από τότε που προσχώρησε το 2011. Και υπάρχουν και αυτά αποτελέσματα από το τι έγινε με, τις, μετρακοστάσια κονσερβοποίησης του τόνου, α πούμε. Κονσερβοποιημένου τόνου ε, εκατοντάδε χιλιάδε θέσει εργασία, ιδίω για τι γυναίκε τη χώρα. Τώρα διερευνούμε με του εταίρου μα πώ μπορούμε να επαναλάβουμε αυτή την επιτυχία των κονσερβών τόνου και σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείε και σε άλλα μέρη του ειρηνικού κοντά στην Νέα Γουινέα. Για μας λοιπόν είναι απλώς λογικό να θέλει και η Σαμόα να υποφεληθεί. Η συμφωνία πλαίσιο για αυτή τη συμφωνία είναι η συμφωνία της Κοτονού. Ε, κεντρικό σημείο είναι η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά μέτρα που θα πρέπει να προβλεφθούν, να ε, ενεργοποιηθούν να υπάρξουν παραβιάσεις. Αυτό είναι κάτι που σκοπεύει να το εξακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάδοχο συμφωνία. Υπάρχει λοιπόν μια πραγματική ακολουθία ε, στις διάφορες συμφωνίες μεταξύ τους, διότι η συμφωνία μετά την, για τη φάση μετά την θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σε ένα χρόνο από τώρα. Ευχαριστώ, David. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για τις απαντήσεις της. Το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι ότι εδώ δεν προσπαθούμε να τιμωρήσουμε ή να στριμώξουμε τους ε, Σαμοέζους. Είναι μια λιγότερα αναπτυγμένη χώρα Δεν λέμε ότι αυτό θα το αλλάξουμε, απλώς Μόνο η εγώ είναι και τα Φίτζι ε, είναι αυτή τη στιγμή ασφαλή λιμένα στον Ειρηνικό. Η Σαμόα θέλει να προσχωρήσει από ό,τι φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει καταλάβει. Γι' αυτό κάνει αυτή την πρόταση. Και δεν βλέπω λόγο να, το λόγο να μην ικανοποιήσουμε το αίτημα της Σαμόας. Οι Σαμοέζοι το ζητάνε. Γιατί να μην του ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ υποβολή για την προθεσμία τροπολογιών 6 Νοεμβρίου. 6 το βράδυ. 6 ε, το βράδυ, 6 Νοεμβρίου. Σημείο 13. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα. Floor immediately. Η συγγήτρια κυρία Λόλα Σάντζεθ έχει το λόγο. Α, θέλετε κάτι άλλο. Ναι, εγώ άκουσα την εκπρόσωπο της Επιτροπής, αλλά δεν μου απάντησε για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του 2018 που εξηγεί ότι μπορούν χωρίς ποσοστός, εκτός ποσοστώσεων να έχουν συναλλαγές δεν ξέρω, αυτό δεν ισχύει στι συμφωνίε με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, έτσι δεν είναι. Απάντησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη που ξέχασα την ερώτησή σας. Πράγματι, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία είναι κύριοι εξαγωγής προϊόντων στη Σαμόα. Όταν διαπραγματευτήκαμε την πρόσβαση στην αγορά με την Σαμόα, αυτό το είχαμε υπόψη μας και τους βοηθήσαμε, γιατί πράγματι δεν ανησυχούν πω πλημμυρίσουν από ευρωπαϊκά προϊόντα γιατί δεν κάνουμε τόσο μεγάλε εξαγωγέ προ τα εκεί. Μηχανήματα, εξοπλισμό εξάγουμε. Ενώ τα προϊόντα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία που βασίζονται στην Συμφωνία Plus όντως ε, κινδυνεύουν να κατακλείσουν τις αγορές μας. Όμως δεν ισχύει ακόμα αυτή η συμφωνία. Έχει μία ρήτρα ασφάλειας που σημαίνει ότι αν η Σαμόα προσχωρήσει στη συμφωνία αργότερα από την από την τότε θα πρέπει ορισμοί να επεκταθούν και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τώρα όμως Είμαστε ένα βήμα πιο πέρα. Και είπα θα αρχίσει να ισχύει πριν από το PESI Plus με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Υπάρχει αποκλεισμό προϊόντων που το λαμβάνει υπόψη. Αν ε, τα πράγματα καταλήξουν ε, με διαφορετική σειρά, θα προστατεύεται η Σαμόα γιατί έχει αποκλείσει προϊόντα τα οποία παράγονται και εισάγονται από τη Νέα ε, Ζηλανδία και την Αυστραλία. Ωραία, ευχαριστούμε. Πάμε πάλι ιατρικά ακόμα. Φάρμακα, η κυρία Λόλα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω λιγάκι για αυτά τα πιστοποιητικά συμπληρωματικής προστασίας. είναι κάτι που πάει πιο πέρα από την νομοθετική πρόταση. Οι οργανώσει ασθενών και όσοι εργάζονται στον κλάδο που σώζουν ζωές προσέχουν τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Στο όνομά τους λοιπόν και στο όνομα τη υγεία τους θέλω να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η επέκταση ε, πατέντας των φαρμάκων. Δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνει περήφανη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μας στοιχίζει σε υγεία αλλά και σε ανθρώπινες ζωές. Μην ξεχνάμε ότι η πρόταση αυτή τροποποίησης του κανονισμού SPC έρχεται σε μια ιστορική στιγμή. Κάποιες χώρες περνάνε από πολύ σοβαρές δυσκολίες για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε φάρμακα των πολιτών. Οπότε η ομάδα μας θα ήθελε σήμερα να μην καθίσουμε και να σκεφτούμε μόνο πώς να βλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συμφωνίες αυτές τύπου SPC, αλλά να δούμε πώς θα έχουμε μια ρύθμιση που δεν θα ζημιώνει την κοινωνία, που θα προσφέρει ωφέλη. Κάτι το οποίο σήμερα είναι πολύ αμφίβολο. Τώρα, πιο ρεαλιστικά. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος και ελπίζω να συνεργαστούν όλοι οι σκιώδες συζητητές σε αυτήν την έκθεση στην οποία ελπίζω να πετύχουμε ε, ευρεία συμφωνία. Υπάρχει αυτή η πρόταση λοιπόν τη Επιτροπής που όντως αμβλύνει κάποιε από τι αρνητικέ επιπτώσει τη συμφωνία SPC. Παρ' όλα αυτά όμω, έπαξε και έχει εντοπιστεί το ζήτημα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε στα μέσα του δρόμου και πρέπει να δούμε και άλλες επιτυχίες που έχει αυτή η πρόταση. Συνεπώς, προτείνω ένα βήμα παραπάνω σε τρεις πολύ συγκεκριμένες πτυχές. Πρώτον, για την είσοδο στην αγορά εργασίας, όταν σταματάει να ισχύει το SPC. Προτείνει η Επιτροπή δύο κλάδους από τους οποίους μπορεί να υπάρχουν ωφέλη. Πρώτον, να υπάρχει ένα διαφορετικό προφίλ των επιχειρήσεων και των παρασκευαστών της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης. Και δεύτερον, να υπάρχουν ωφέλη για τους ε, Ευρωπαίους ασθενούς, ασθενείς. Και οι δύο αυτές στόχοι, ο δεύτερος κυρίως, δεν ολοκληρώνεται αν δεν υπάρχει δυνατότητα. Μία επιχείρηση η οποία παράγει για νόσημα και βιομηδή φάρμακα ε, δεν θα είναι σε θέση να ε, εισάγει τα προϊόντα της στην ευρωπαϊκή αγορά όταν ε, εκπίπτει το SPC. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το απαιτήσουμε. Δεύτερον, πώς εφαρμόζονται τα μέτρα του ισχύοντο SPC. Για να υπάρχει μια πραγματική επίπτωση, δεν φτάνει η εξαίρεση να εφαρμόζεται μόνο στι συμφωνίε SPC που δεν ισχύουν ακόμα. Πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε του λογαριασμού μα. Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να περιμένουμε πέντε χρόνια τουλάχιστον ή και παραπάνω για να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Οπότε, τι γίνεται με τον μεγάλο αριθμό ασθενών ε, τα επόμενα χρόνια όταν θα έχουν εκπέσει αυτές οι συμφωνίες. Πώς θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις. Για πέντε χρόνια δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι η εξαίρεση αυτή δεν ε, αφαιρεί κανένα δικαίωμα από τις εταιρείες που παράγουν αυτά τα φάρμακα. Μόνο όταν εκπνέει συμφωνία σπίση οποιαδήποτε επιχείρηση από οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε αν μη τι άλλο και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν το ίδιο. Έπειτα για θέματα διαφάνειας και σήμανσης πρέπει να υπάρχει μια ειδική ετικέτα μόνο για εξαγωγή, είπαμε, για να μην γίνονται παράνομα επανεισαγωγές. Αυτό είναι κατανοητό ως φόβος, αλλά πρέπει να αποφύγουμε να παίρνουμε και λάθος αποφάσεις βασισμένοι ακριβώς σε αυτό. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το ότι έχουμε ένα σύστημα ανείχνευσης των πλαστών φαρμάκων που λειτουργεί και αποτελεσματικά. Ζούμε σε έναν κόσμο που η τεχνολογία μας επιτρέπει να είμαστε σίγουροι για την προέλευση των φαρμάκων που καταπίνουμε, χωρίς να χρειάζεται μια παραπάνω σφραγίδα στο πακέτο. Το μόνο, και το μόνο που θα έκανε μια από πάνω ετικέτα είναι ότι θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα στις πιο μικρές επιχειρήσεις παρασκευής φαρμάκων. Πρέπει να διευκολύνουμε μια επιχείρηση που θέλει να χρησιμοποιήσει την εξαίρεση. Γι' αυτό πρέπει οι υγειονομικές αρχές να έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η προστασία των πολιτών. Και αν δεν πρόκειται μόνο για αυτό, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα αποκαλύπτονται εμπορικά στοιχεία για τις εξαγωγές και για την ημερομηνία που θα γίνει η εξαγωγή. Το να αποκαλύπτουμε πληροφορίες, αυτό κοστίζει στις επιχειρήσεις παραγωγής γενώσιμων προϊόντων και δεν προσφέρει κανένα όφελο στο κράτος ή στους πολίτες. Το να επιβάλλουμε στις ε, επιχειρήσεις που παράγουν φάρμακα πράγματα τα οποία οι υπόλοιπες εταιρείες δεν θα δεχόντουσαν με τίποτα, ε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισόρροπο παιχνίδι εδώ και δίκαιο. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να πετύχουμε μια συνένεση μεταξύ όλων των ομάδων. Ευχαριστούμε κύριο Σχέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά παίζω το ρόλο του Ντάνιελ Γκάσπαρη αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, επειδή προερχόμαστε από διαφορετικές οπτικές γωνίες ο καθένας μας αυτή τη συζήτηση, από ό,τι ξέρω τα νέα καινοτόμα φάρμακα δεν πέφτουν από τον ουρανό με τη βροχή, κάποιος τις παράγει με μια συγκεκριμένη διαδικασία και εμείς σαν πολιτικοί, αλλά και σαν ασθενείς ενδεχομένως, Θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν αυτά τα ε, φάρμακα και φυσικά χωρίς ε, την προστασία αυτής της καινοτομίας δεν μπορούν να υπάρξουν νέα φάρμακα. Τα SPC άρχισαν να ισχύουν ακριβώς επειδή ο χρόνος προστασίας γινόταν όλο και πιο σύντομος διότι η διαδικασία έγκρισης και άδεια για να μπει ένα φάρμακο στην αγορά γινόταν όλο και πιο δύσκολη και όλο και πιο χρονοβόρα. Η πρόκληση της ε, Επιτροπής, αν θέλετε, είναι να βρεθεί μια ισορροπημένη θέση μεταξύ του να μην υπονομεύσουμε ε, την καινοτομία, τη δυνατότητα παραγωγής νέων καινοτόμων φαρμάκων που χρειάζεται όχι μόνο η Ευρώπη αλλά ο κόσμος και η, ο κλάδος των ε, γενοσύμων να μπορούν να επιβιώσουν και να εξάγουν σε χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα φάρμακα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να παραμείνουμε κοντά στην παρακολούθηση που έχει κάνει μέχρι σήμερα η Επιτροπή. Η προσέγγιση του εισηγητή πιστεύουμε ότι είναι πολύ κοντά στην, στον κλάδο των γενοσύμων. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι αν δεν υπάρχουν πρωτότυπα και καινοτόμα φάρμακα, δεν υπάρχουν γενόσημα. Είναι λοιπόν αλληλοεξαρτώμενοι αυτοί οι δύο τομείς. Γι' αυτό και θα ήθελα να επανέλθω στην Επιτροπή. Και θα κάνω μία ερώτηση προς την Επιτροπή πριν ολοκληρώσω. Τα SPCs δεν είναι απλώς ένα πολύ σημαντικό τμήμα των δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων και της προστασίας των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μεταρρύθμιση αυτή καταλαβαίνει η Επιτροπή ότι μπορεί να υπονομεύσουμε άλλες διαδικασίες SPC σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Η Αλέσια Μόσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι είναι μια καλή πρόταση και θα μπορούσε να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια σημεία, κάποια στοιχεία της πρότασης αυτής. Καταρχήν να πω ότι πιστεύουμε ότι ο αρχικός σκοπός είναι να υπάρχει αξία, να εγγυηθούμε την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο και πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην υπόσχεση του Επιτρόπου όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στις επιπτώσεις επί των πολιτών. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Η πρόταση αυτή σίγουρα δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή γενώσιμων και βιοπαρόμοιων φαρμάκων καθότι θεωρούμε ότι πρέπει αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στα ακριβότερα φάρμακα να μπορούν να επωφεληθούν από την παραγωγή αυτή. Και ενώ εμείς ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό στον τομέα αυτό, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν πρακτικές ε, οι οποίες δεν είναι αθέμητες στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Τρίτον, πολύ σημαντικό να δούμε και τις ε, επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να λάβουμε υπόψη μας και τα τρία αυτά σημεία. Συμφωνώ με τις προτάσεις αυτές οι οποίες ε, αποσκοπούν στο να βρεθεί αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχουν κάποιες τροποποίησεις ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα των ε, του waiver, το πού μπορεί να εφαρμοστεί, υπό ποιες προϋποθέσεις και το θέμα του να δίνονται απαραίτητες ε, πληροφορίες ε, σε αυτούς οι οποίοι είναι κάτοχοι SPC, αρκετές έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν την ίδια ώρα και τα γενώσιμα και βιοπαρόμοια φάρμακα. Οι κάτοχοι SPC θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο. Ολοκληρώνω και θεωρώ ότι ένα καθοριστικό τμήμα αυτού του κανονισμού είναι ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην αγορά από την πρώτη μέρα, να δημιουργούμε δηλαδή κατάλληλες συνθήκες στην αγορά για να μπορούν να επιβιώσουν τα φάρμακα αυτά. Γι' αυτό και το θέμα του waiver σε υπάρχοντα SPC θα πρέπει να είναι προκαθορισμένο καθώς και οι όροι της ισχύω του. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτές μας οι προτάσεις να έχουν θετικές επιπτώσεις και στους πολίτες αλλά και τις θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η φαρμακοβιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να περάσει ανταγωνισμό με τους παραγωγούς γενοσύμων και δύο αντιστοίχων, όπως ονομάστηκαν. Δεν θα πρέπει αυτούς να τους περιορίσουμε θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως το ε, δυναμικό τους, γιατί υπάρχουν και παραγωγή των τρίτων κρατών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσει το 2020, θα έχουμε ένα σωρό διπλώματα ευρεσιτεχνία που θα εκπνεύσουν για φάρμακα αξίας 90 δις ευρώ. Η φαρμακοβιομηχανία λοιπόν θα πρέπει να μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε αυτή την αγορά. Σήμερα όμως υπάρχουν πολύ περιοριστικές ε, ρυθμίσεις. Φυσικά χρειάζονται μέτρα προστασίας για να μην υπάρχουν ανεξέλεγκτες ε, εξαγωγές προς το εξωτερικό πρώτα και μετά προς τα άλλα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, πρέπει να επιτρέψουμε και στις ευρωπαϊκές εταιρείε να αναπτυχθούν γιατί οι υπόλοιπε εταιρείε της Κίνας και άλλων περιοχών δεν δίνουν σημασία σε αυτά. Στηρίζουμε λοιπόν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμη και αν έχουμε αρκετούς ενδιασμούς ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, επιβολή των μέτρων αυτών στην ε, σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Θα πρέπει να δούμε σε ποια θα επιβληθεί. Και θέλουμε ο κανονισμό να ωφελήσει πραγματικά τις εταιρείε, ιδίως τις μικρομεσαίες. Θα υποβάλουμε τις σχετικέ τροπολογίες και υπολογίζουμε στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά τα βιολογικά αντίστοιχα, τα γενώσιμα φάρμακα και να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της βιομηχανίας των γενώσιμων και του υπόλοιπου ε, κομματιού της βιομηχανίας. Ευχαριστούμε. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πρότασή του μια-δυο παρατηρήσεις από την πλευρά μου. για την καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα. Ο βασικός στόχος της πρότασης αυτής είναι μια ε, στρατηγική για την ε, ενιαία αγορά και για να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας. Βεβαίως, εάν προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο και στην πρόσβαση στα φάρμακα κάτι που εξηγείται πολύ καλά στην ε, πρόταση, στην έκθεσή σας. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με την έκθεση είναι η Ευρωπαίοι παραγωγοί σε νέε αγορέ για γενοσύμα και αντίστοιχα να πετύχουν να είναι ανταγωνιστικοί. Ω τώρα, ευρωπαϊκέ εταιρείε επενδύουν στην Ευρώπη. Επενδύουν στην Ευρώπη με σκοπό να εξάγουν σε τρίτε χώρε, ακόμη και κατά την ε, φάση του SPC. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι οι δικοί μα, οι Ευρωπαίοι ασθενεί, έχουν πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Ιδίω μετά την εκπνοή της προστασίας Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε την συνέχεια που θα δοθεί στο σύστημα SPC. Επίσης, τη χρονική εφαρμογή. Μόλις εξήγησα ποια είναι η δική μας άποψη, βεβαίως είμαστε υπέρ της ταχείας της εφαρμογή του waiver της εξαίρεση. Αλλά πρέπει να δούμε ότι γίνονται και τα πράγματα σωστά. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των εξαιρέσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τις εγγύησεις, ακούω κάποιες προτάσεις από τα μέλη της Επιτροπής σας. Δικός μας στόχος ήταν να κάνουμε μια πρόταση που να καλύπτουν στο δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Προσθέσαμε κάποια πράγματα γιατί αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις όπου φάρμακα παρασκευάζονται στην Ευρώπη και θα έχει ακόμα η προστασία SPC. Γι' αυτό χρειάζονται αυτά τα τμήματα ώστε να αποφύγουμε την παρανομή, τις παρανομίες και τις στην ευρωπαϊκή αγορά για αυτό το διάστημα. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι διασφαλίσεις δεν πρέπει να γίνουν επαχθείς δεν πρέπει να προσθέσουν φόρτο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ισορροπημένη η πρότασή σας, αλλά καταγράφουμε και τις προτάσεις σας με προσοχή. Θέλουμε να, υπάρχει η να υπάρχουν σωστές διασφαλίσεις, όπως ας πούμε ο μοναδικός ε, υπεύθυνος για την ταυτοποίηση. Και για το θέμα που τέθηκε από τον κύριο Φιέλνερ και πώς η πρότασή μας αυτή ε, συνδυάζεται με τις προσπάθειές μας στο επίπεδο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Όντως, η πρότασή μας με την εξαίρεση για τις εξαγωγές συνάδει πλήρως με τις προσπάθειές μας για να έχουμε τη σωστή προστασία σε διεθνές επίπεδο. Το κάναμε ανέκαθεν, συνεχίζουμε Είχαμε και την πρόσφατη συμφωνία με τον Καναδά, όπου είχαμε το τέτοιο σύστημα SPC, με εξαίρεση για τις εξαγωγές Και όταν συνεχίσουν να υπάρχουν αποκλήσει, θέλουμε οι ευρωπαϊκέ εταιρείε να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Δηλαδή, θέλουμε οι εταιρείε μα να ανταγωνίζονται με ίσου κανόνε και όρου παιχνιδιού στη διεθνή αγορά και το επίπεδο προστασία να αυξηθεί παγκοσμίω. Να υπάρχει απόλυτη συμπληρωματικότητα, να κουμπώνουν τα δύο επίπεδα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σάντσε. Ευχαριστώ κάποια σχόλια και διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν λέμε ούτε η ομάδα, ούτε εγώ σε συγκίτρια, ούτε η Επιτροπή αυτή, να περιορίσουμε τα δικαιώματα του επενδυτή που προβλέπει το SPC γεωγραφικά. Ισχύει το SPC στο διάστημα που ισχύει και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτό που λέμε είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δρούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες όπως και οι τρίτες χώρες μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά, άπαξ και έχει εκπνεύσει το SPC. Δεύτερον, στόχος της πρότασης αυτής είναι να μην υπάρχουν πια τα αρνητικά από την εισαγωγή της συμφωνία SPC. Άπαξ και ισχύσει, κανείς δεν μπορεί να πουλήσει στην Ευρώπη ούτε στο εξωτερικό. Όμως επιχειρήσεις που έχουν τη βάση τους εκτός Ευρώπης μπορούν να κάνουν τέτοιες εξαγωγές προς χώρες που δεν έχουν τις εξαιρέσεις. Οπότε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις των γενώσιμων φαρμάκων δεν θα πρέπει να πηγαίνουν αλλού, θα πρέπει να μπορούν να μένουν μέσα και να μπορούν όμως να κάνουν αυτό τον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπε. Αλλιώς χάνουν πολλά. Αυτές που είναι στο εξωτερικό μπορούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη μέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε έκθεση στο, σαν Ινστιτούτο Οικονομικών που λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιο κομμάτι των χρημάτων που προσφέρεται στις επιχειρήσεις μέσω φόρων και λόγω του μονοπωλίου επανεπενδύεται. Γιατί τα στοιχεία δεν βοηθούν, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την απόσβεση της ε, επένδυσης πόσα από τα χρήματα αυτά επιστρέφουν, άρα να βγάλουμε το συμπέρασμα πόσο χρήσιμο είναι το SPC ή δεν είναι. Αν δεν έχουμε στοιχεία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Τέλος. Με την εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων θα είμαστε σίγουροι ότι είμαστε συνεπείς υπέρ της ανάπτυξης. Ότι δηλαδή δεν δυσκολεύουμε υποανάπτυξη χώρες προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους φαρμακευτικές βιομηχανίες. Αυτά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 7 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίας. 6 μετά μεσημβρίας. Ευχαριστούμε. Αυτό εδώ το σημείο 13 και περνάμε στο σημείο 14. Πρόκειται για θέσπιση μηχανισμού προενταξιακή βοήθειας. Η συγητή είναι ο κύριος Μπορέλη. Παρακαλώ, κύριε Μπορέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση κανονισμού ε Τη οποία ε, εγκύπτουμε ε, ε, ασχολείται με την τοποθέτησή μα για ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα για το μέλλον τη Ευρώπη. Τη δυνατότητά μα να ανεχθούμε σε νέε χώρε, προσπαθώντα να εδραιώσουμε και τι δικέ του θεμελιώδει αξίε. Γι' αυτό το λόγο η γνωμοδότησή μας δεν μπορεί να αποφύγει δύο βασικά σημεία από τα οποία ξεκινεί ξεκινά η εξέταση του θέματος. Οι υποψήφιε χώρε αυτή τη στιγμή ε, έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσει γεωπολιτικέ που έχουν αλλάξει πολύ και ε, από τότε που ξεκίνησε την πολιτική διεύρυνση στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η δεύτερη είναι ότι πρέπει να ε, προσαρμοστούμε στι περίπλοκε συνθήκε του παρόντο και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει τον σεβασμό θεμελιωδών αξιών μεταξύ των οποίων αυτών που επηρεάζουν την εμπορική πολιτική. Υπό αυτή την σκοπιά ε, έχει σημασία να επιδιώξουμε ένα οικονομικό εργαλείο υποστήριξη χωρών που θέλουν να ενταχθούν και να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω πρέπει να υπάρξει προσεκτική και διαρκή παρακολούθηση του κατά πόσον ε, η βοήθεια που παρέχεται οδηγεί σε αυτά αποτελέσματα. Υπό την ιδιότητα του εισηγητού σε αυτή την επιτροπή έχω την πρόθεση να ε, τονίσω τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές πτυχές της στρατηγικής της Ευρώπης για τη διεύρυνση και θέλω να σταθώ σε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα. Πιο συγκεκριμένα την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραποίησης, ε, της πειρατείας. Θα πρέπει να παραμείνουν μια θετική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εμπορικές συναλλαγές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χώρες. Παρά τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει, οι συναλλαγές που είναι παράνομες γραμμές αυξάνονται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πιο αποφασιστική αντίδραση στο επίπεδο της τελωνιακής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Επιπλέον, γραμμή που καθοδήγησε τις ε, εμπορικές μας σχέσεις ε, με τις τρίτες χώρες, ιδίως τις υποψήφιες για την ένταξη, είναι η θέσπιση ενός ανοιχτόμυαλου εμπορικού πλαισίου που να βασίζεται σε σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες. Όμως, την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους φραγμούς ε, ει βάρο του εμπορίου και των επενδύσεων, η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν ανατρέξει ω περισσότερο από άλλε μέτρα προστατευτισμού και εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε απομακρύνονται από τη συμφωνία που ισχύει για την Τελωνιακή Ένωση. Εάν λοιπόν αξιολογήσουμε τι προσπάθειε που κάνουν οι χώρε αυτέ, έχοντα επίγνωση ότι σημαντικά βήματα προόδου γίνονται στον τομέα τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, Οπότε ε, σίγουρα εδώ πέρα κάπως αντιμετωπίζεται και το παράνομο εμπόριο. Πρέπει να προστατευτούν και οι ξένες επενδύσεις και οι εμπορικές συναλλαγές μέσω της άρσης των ανεπιθύμητων και αδικαιολόγητων δασμών και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η πρώτη εκδοχή της ε, γνωμοδότησης να εμπλουτιστεί και να ε, προσαρμοστεί στις επιθυμίες των συναδέλφων με τις συνασφορές τους. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ το χρήμα. Η S&D. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Χάνζεν, πριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι εδώ στη θέση της κυρίας Αντρίκεν, που είναι η σκιώδη συγγήτρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσει καταρχήν τον εισηγητή, μέρος της ΣΥΝΤΑ, για την εξαιρετική μέχρι τώρα εργασία. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε περισσότερη σταθερότητα, ασφάλεια αλλά και βιώσιμη οικονομική ανάκτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα μελλοντικά σημεία επένδυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερη ευημερία για τις γειτονικές μας χώρα. Η διεύρυνση αυτής της πολιτικής σίγουρα θα βοηθήσει σε καλύτερες συμφωνίες και πιο ελεύθερη και ανοιχτή πολιτική στον τομέα των συναλλαγών. Θα πρέπει επίσης να προστατεύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την λειτουργία της οικονομίας της αγοράς με βελτιωμένους κανονισμούς και με επενδύσεις που θα στηρίζουν τη βιώσιμη οικονομία. Η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς είναι καθοριστικός παράγοντας για να προσελκύσουμε νέους επενδυτές. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα, θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή όλων όσον αφορά την τήρηση των αρχών, των συστημάτων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει τα εργαλεία αυτά να βοηθούν αυτούς που θέλουν να επενδύσουν σε ξένες χώρες της Βαλτικής βαλκανικές χώρες, την Τουρκία, έτσι ώστε να στηρίξουν την οικονομία αυτών των χωρών με κανόνες ε, δίκαιου ανταγωνισμού και σεβασμό των ε, ρυθμίσεων. Θα πρέπει την ίδια ώρα να, ισχύσει η, να ισχύσουν οι προτεραιότητες, οι όροι, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία Αυτές είναι οι κύριες ιδέες ε, της κυρίας ε, Αντρέκινεν και η οποία μου ζήτησε να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος του κυρίου Κώστα Μαυρίδη. Καταρχήν ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έξισης. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος και πολύ σύντομος. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να στηρίξουμε οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις σε χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για κάτι που συμβαδίζει με την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέλουμε να διασφαλίσουμε ίση κατανομή στις διάφορες περιοχές και μια ισορροπημένη προσέγγιση έτσι ώστε όλοι οι πολίτες από όλες τις κατηγορίες τις κοινωνικές να επωφεληθούν από αυτές τις νέες διατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις και βεβαίως το σεβασμό των, ε, της κοινωνικής διάστασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης για όλη την διανομή και κατανομή των πόρων. Θέλουμε επίσης να δούμε και μία πιο ισχυρή κοινωνική διάσταση κατά την διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια παρακολούθηση όσον αφορά την κατανομή των πόρων και στις ε, χώρες αυτές καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν ε, επικοδομητικές ε, και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα σε αυτή την έκθεση, γιατί κάποια σημεία που προστίθενται φαίνεται να έχουν ε, εξαφανιστεί. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω και βρίσκομαι σε σύγχυση. Επίσης υπάρχουν πολλά σχόλια που είναι ιταλικά. Εγώ όπως και άλλοι φαντάζομαι δεν είμαι γνώστης της ιταλικής γλώσσας. Σας παρακαλώ ελπίζω τα τεχνικά σημεία που θα προσθεθούν να γίνει ε, αυτό με μεγάλη προσοχή. Τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα και έχουν απόλυτη σχέση με θέματα Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών και Ανάπτυξης των χωρών αυτών. Η πρόσβαση αγορές για τις χώρες αυτές θα πρέπει να επιτευχθεί με την εναρμόνιση και συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας με το κοινοτικό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια πολιτική εμπορικών συναλλαγών με μας. Αυτό κάπου σε κάποια τροπολογία θα πρέπει να αναφερθεί. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η φιλελευθερωποίηση των ε, συναλλαγών, οι συμφωνίες σύνδεσης, αλλά και άλλου είδους ασυμμετρικές και σταδιακές ε, συμφωνίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν ε, πλήγματα για τις ευαίσθητες αυτές οικονομίες. Όσον αφορά την Τουρκία, πιστεύουμε ότι οι οικονομικές μας σχέσεις αλλά και οι άλλες σχέσεις με τη χώρα αυτή θα πρέπει να συζητηθούν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και όχι εδώ ε, σε αυτό το συγκεκριμένο που συζητούμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Thank you. για την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα πλαίσιο για το θέμα των δασμών, η ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά σημεία. Θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε μία από τις τροπολογίες, την 9, που αναφέρεται στο γεγονός ότι η οικονομική πόρη από το ΙΠΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο και εφόσον εάν προοδεύουν προς τους ευκταίους στόχους και επίπεδα όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα 1 Ήθελα να πω ότι σκοπός μας είναι να μην υπάρχουν πλέον ε, συνολικά ποσά αναχώρα και να στοχεύσουμε σε επιδόσεις. Δηλαδή σε σχήματα χρηματοδότησης που θα βασίζονται σε μετρήσεις των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας. Θεωρούμε ότι οι στόχοι του ΙΠΑ θα πρέπει να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να φτάσουν στους στόχους αυτούς και να μην θεωρηθεί ότι είναι προϋπόθεση η επίτευξη των στόχων αυτών για να δοθεί η βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μπορέλη. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις τους. Ήταν η πρώτη συζήτηση που κάναμε από το θέμα τους, οπότε θα κοιτάξουμε να διοργανωθούμε και για τα τεχνικά θέματα και για τις μεταφράσεις και για την πολιτική διάσταση του θέματος με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. So deadline for tabling Ευχαριστούμε. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 8 Νοεμβρίου, 6 το απόγευμα, δηλαδή 6 που μου, 8 Νοεμβρίου. Μου μου μάλλον. Ε, ολοκληρώσαμε το σημείο 14 και τώρα περνάμε στο 15, 16 και 17 που θα τα εκτάσουμε από κοινού. Έρχεται ο εισηγητή και θα κάνω ένα διάλειμμα λεπτό. Ένα λεπτό. Εντάξει, παιδιά, δεν πάω καλά. Okay. Dear colleagues. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, 15, 16, 17. Πρόκειται για την αντιπροσωπεία μας στη Δυτική Σαχάρα και την συμφωνία υπό την μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου. Η συγκίτρια για όλα αυτά τα θέματα είναι η κυρία Λαλόντο. Οπότε, της δίνω το λόγο για 4-5 λεπτά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω από κοινού να εξετάσω αυτά τα τρία θέματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο ζήτημα, συνδέονται μεταξύ τους. Τον ε, Ιούλιο ζητήθηκε από το κοινοβούλιο μας να επικυρώσει όχι τη συμφωνία αυτή. Πρόκειται για μια συμφωνία κάπως ε, διαφορετική, γιατί υπήρχε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έκρινε ότι η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου δεν ήταν εφαρμόσιμη ως είχε στην επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας. Για το δικαστήριο Πρέπει να υπάρχουν δύο προποθέσει. Πρώτον, να αναφέρεται ρητά η επικράτεια της Δυτική Σαχάρας στο κείμενο και δεύτερον, να έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη του πληθυσμού της Σαχάρα. Οπότε εδώ πέρα βασιζόμαστε στη Σύμβαση της Βιέννη. Και υπάρχει λοιπόν ένα επιπλέον κριτήριο που είναι εκείνο του ωφέλους για τον τοπικό πληθυσμό. Και βάσει αυτών των τριών στοιχείων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε την τροποποιημένη συμφωνία πάνω στην οποία πρέπει να αποφαθούμε με σήμερα. Η μέθοδος εργασίας που ακολουθήσαμε ήταν να συλλέξουμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τους ίδιους μέσω συναντήσεων με τα διαφερόμενα μέρη. Και έτσι λοιπόν είχαμε ανταλλαγέ απόψεων με την κοινωνία των πολιτών, τους τοπικά εκλεγμένους και το μέτωπο Πολυσάριο. Επίσης, πήγαμε επί τόπου σε μία αποστολή fact-finding, όπως τη λέμε, διερευνητική, όπου πέντε διαφορετικές πολιτικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Τελικά κατέληξαμε σε τρεις πολιτικές διαφορετικές ομάδες. Η διάσκεψη των Πρόεδρων μας επέτρεψε για δύο μέρες να πάμε στη Δυτική Σαχάρα. Το τμήμα εκείνο δηλαδή που καλύπτεται από τις προτιμησιακές συμφωνίες ε, στις οποίες αναφέρεται το δικαστήριο. Πήγαμε λοιπόν και προσπαθήσαμε να συναντηθούμε όσο γίνεται περισσότερους φορείς από διάφορα τμήματα της κοινωνίας για να ε, δημιουργήσουμε μια πλήρη εικόνα. Άκουσα δεξιά και αριστερά σχόλια που λέγανε ότι δεν ήταν ισορροπημένη η αντιπροσωπεία μα, ότι δεν συναντηθήκαμε με αρκετού φορεί από την κοινωνία των πολιτών κτλ. Η απάντησή μου είναι ότι συντονιστήκαμε με διάφορε ομάδε τη κοινωνία των πολιτών επιτόπου, ότι ήμασταν στη διάθεση των αντιπροσώπων του για να του ε, δούμε και να του ακούσουμε. Οπότε υπήρχαν κάποιοι που ήταν υπέρ του Μαρόκου, κάποιοι που ήταν ουδέτεροι αλλά θέλανε καλύτερε συνθήκε παραγωγή ε, ή απλώ ήταν υπέρ του Παλισόρου. Εγώ δεν είμαι αφελή και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν όλοι να συμφωνήσουν στην αντιπροσωπεία μα γιατί ξέρω και τι διακυδεύεται. Όμω πρέπει να σα διαβεβαιώσω ότι δούλεψαμε σκληρά ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε κάτω από τι συγκεκριμένε συνθήκε. Συναντηθήκαμε λοιπόν με διάφορου φορεί, με οικονομικού φορεί οι οποίοι ζουν από τα προϊόντα τα οποία αφορά ακριβώ αυτή η συμφωνία. Και το συμπέρασμά μα είναι πρώτα απ' όλα ότι είναι μοιρασμένε οι απόψει ανάλογα με το πλαίσιο, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιέφερε πάνω απ' όλα ήταν η προτίμηση. Και αυτό που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε είναι να μπορούν από αυτές τις προτιμήσεις να ωφεληθούν οι άνθρωποι που ζουν επί τόπου. Γιατί είναι ένας τρόπος που τους προσφέρει περισσότερη αυτονομία απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση όταν μπορούν απευθείας να εξάγουν σε μας. Είχαμε διάφορες λοιπόν ανταλλαγές απόψεων και να τις σας προτείνω. Πρώτον, η δουλειά γίνεται στα πλαίσια μιας ειρνευτικής διαδικασίας, παράλληλα διότι υπάρχει και ο πρόσωπο του ΙΕ που δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει τα διάφορα μέρη το Δεκέμβριο. Εμεί στηρίζουμε το δικό του το διάβημα και είμαστε τακτικά σε επαφή με του συνεργάτε του. Να το ξέρετε δηλαδή, μπορεί να έχουμε διαφορετικέ αποστολέ, αλλά συντονίζουμε τη δράση μα με τον ΟΗΕ. Και είναι κάτι που το συζητήσαμε και επί τόπου. Δεύτερο, για το νομικό σκέλο. Ε, αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι υπάρχει μια βεβαιότητα. Γι' αυτό και το σχέδιο εκθεσή μα που συνοδεύει τη σύσταση παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτικό για αυτό το σημείο για το θέμα της σύμφωνη γνώμη. Τρίτον, πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν σωστό να τιμωρείται ο τοπικός πληθυσμό από... αφαιρώντας του τις προτιμήσει περιμένοντας μια πολιτική συμφωνία. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν ε, προτιμησιακή ε, πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Τέλος, για όλους αυτούς τους λόγους συστήνω να κυρώσουμε την συμφωνία αλλά υπό προϋποθέσεις που είναι οι εξής. Πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός συγκεκριμένος χρησιμότητα των προϊόντων που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε πολύ συγκεκριμένα ποια προϊόντα εξάγονται από τη Δυτική Σαχάρα και ποια εξάγονται από το υπόλοιπο Μαρόκο. Δεύτερον, η ίχνηλασιμότητα αυτή θα πρέπει να είναι τεχνική φύσεως. Πρέπει να γίνεται αναπροϊόν έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το τι εξάγουμε από τη Δυτική Σαχάρα και έτσι να μην υπάρχει τόσο πολύ νομική βεβαιότητα. Για μένα είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ε, κυρώσουμε τη συμφωνία αυτή. Επίσης πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή και τις επιπτώσεις οικονομικές και άλλες της συμφωνίας, ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά σε συνεργασία με το Κοινοβουλίο μας. Αυτή λοιπόν τη γραμμή υποστηρίζω και σας προτείνω. Να ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι προσβλέπω στις δικές σας προτάσεις και σχόλια. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ε, next. Ευχαριστούμε. Πρώτος σκιώδης εισηγητής ο κύριος Τσίκου από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συγχαρώ την συνάδελφο Εξαιρετική η δουλειά της. Πραγματικά μια ολόκληρη πανδεσία θεμάτων. Κατάφερε να μας δώσει μια παροραμική εικόνα 360 μοιρών το τι γίνεται με τα δικαστήρια, σύγκριση με την τωρινή συμφωνία, όλα αυτά τα στοιχεία που από την ε, πραγματικά νομική σκοπιά, την δικονομική σκοπιά είναι σημαντικά ε, για να μπορούμε να καταλήξουμε σε πραγματική ανασύσταση ε, της εικόνας που χρειαζόμαστε για να καταλήξουμε σε κύρωση. Σε κύρωση που να έχει και κύρος και πρόπτικη για το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εδώ ε, το στοιχείο αυτό το έχουμε εκτιμήσει και έχουμε περάσει στη φάση της αποτίμησης αλλά έχουμε δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε και το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, του ρόλου μας. Δεν μπορούμε εμείς ε, να αναγνωρίσουμε ή να δικάσουμε κανέναν με τη ζυγαριά της Θέμηδος. Η Επιτροπή ε, η ΙΝΤΑ έχει άλλο στόχο και άλλο ε, αντικείμενο. Μιλάμε για εμπορικέ συμφωνίε και κύριο εμπορικών συμφωνιών. Θεωρώ λοιπόν ότι ω προ την κατεύθυνση αυτή και κυρίω την επαλήθευση και τον έλεγχο των ε, ωφελών που μπορούν να προκύψουν για τους πολίτε της Αχάρας. το κατά πόσον τα προϊόντα που εξάγονται είναι αναγνωρίσιμα, το γεγονό ότι θα πρέπει να είναι σαφή πληροφορία για την προέλευση, την καταγωγή αυτών των αγαθών, θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να επιτρέπει ε, να ε, εκπληρώνεται ένα από τα στοιχεία που ανέφερε και το δικαστήριο. Αυτό μου φαίνεται ότι έχει να κάνει και με την πλήρη ε, προθυμία της κυβέρνησης του Μαρόκου να τα υλοποιήσει όλα αυτά και να επιτευχθεί ο συγκεκριμένο στόχο. Ό,τι με αφορά λοιπόν, η θέση μου είναι θετική. Με αυτέ τι διευκρινήσει που έκανα, ίσω να μην υπάρχει πλήρη χνηλασιμότητα, απλώ συγκεκριμένη ενημέρωση ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε την προέλευση του προϊόντος ε, από, που έρχεται από την ε, Σαχάρα. Ευχαριστούμε κυρία Βαλενθιάνο για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο εκ μέρου εμού της ιδίας. Ξέρουν οι υπόλοιποι σχεδόν ότι αυτή τη συμφωνία θέλουμε να την απορρίψουμε. Καταρχάς όμως, όταν λάβαμε την απόφαση του δικαστηρίου για το θέμα, είδαμε αρχικά να υπάρχει μια σειρά από προβλήματα με πρώτο την απάτη. Από την πλευρά της ομάδας μου θέλω να υπάρχει κάποια σύσταση για την μορφή της συμφωνίας και συμπεριζόμαστε το σχέδιο της νομοδότησης και το πνεύμα. Και Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είναι λειτουργικό το, το πλαίσιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν μεταρρυθμίσει ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει η συμφωνία. Η ομάδα μου γνωρίζει τι δυσκολίε ε, που υπάρχουν με τι διαπραγματεύσει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Όμω η πολιτική ασφάλεια και η τεχνική ε, σταθερότητα ε, δείχνει ότι πρέπει να ε, προχωρήσουμε με τη συμφωνία αυτή. Θέλουμε λοιπόν τη μέγιστη συνεργασία και ε, πρέπει να έχουμε αυτό το είδος τη συνεργασία ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προσέξουμε και τη γλώσσα του ψηφίσματος, ώστε να είμαστε αρκετά αυστηροί και να γίνουν σεβαστοί οι όροι μας. Θα πρέπει να, λάβουμε, ε, να ληφθεί σοβαρά υπόψη η άποψη αυτού του Κοινοβουλίου και τα όσα λένε οι βουλευτές αυτού του σώματος. Τέλος, το ψήφισμα θέτει τους απαραίτητες προϋποθέσεις για, ε, για να μπορέσει να απηχηθεί η, η απόφαση του δικαστηρίου στην συμφωνία. Είναι αλήθεια επίσης ότι το ψήφισμα πρέπει να αναφέρεται στα δικαιώματα και στις επιθυμίες του ντόπιου πληθυσμού και στους φορείς της περιοχής αυτής, η οποία έτσι καλλιώς βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών διαδικασιών ιδιαίτερα περίπλοκων και που κρατάνε και πάρα πολύ. Πρέπει όλοι να μπορούμε να δούμε τα θετικά αυτού του μηχανισμού συνεργασίας με μια από τις πιο κοντινές μας γείτονες χώρες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. E Ευχαριστώ για το ECR, κύριος Λούνες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, κυρίως ο συνάδελφος του ΕΛΚ. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πρώτα απ' όλα για την παρουσίασή της. Εμείς θεωρούμε ότι το κείμενο στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι ένα ισορροπημένο κείμενο. Υπάρχει αυτή η διτή προσέγγιση που προτείνουμε. Δηλαδή ότι από τη μια λέμε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και να εγκριθεί η συμφωνία και να προχωρήσει. Από την άλλη μεριά να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον μηχανισμό ο οποίος τεχνικά θα εντοπίζει την προέλευση των προϊόντων που εξάγονται στην Ευρώπη από την περιοχή για να ξέρουμε ποια είναι τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και ποια όχι. Το στηρίζει λοιπόν αυτό και η ομάδα μας. Όπως επίσης και τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΙΕ θέλουμε και εμείς να βρεθεί μια λύση βάσει του διεθνούς δικαίου. Σίγουρα είμαστε ανοιχτοί για παρετέρω καρποφόρα συνεργασία και επικοδομητική με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους ε, σκιώδες εισηγητές πάνω σε αυτό το κείμενο που όπως σας είπα θεωρώ ότι είναι ισορροπημένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε ομάδες που δεν εκπροσωπούνται καν για το θέμα το οποίο ουσιαστικά συζητούμε. Θα ήθελα να πω ότι εκπλήσωμαι πραγματικά γιατί κανείς δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτή η αποστολή και η έκθεση αυτή έχουν ένα εξαιρετικά λεπτό χαρακτήρα και πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το 2016 η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην μη αναγνώριση από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κυριαρχίας του Μαρόκου Σακάρα. Αυτό είναι το σημείο κίνησης και σαν Επιτροπή Ίντα βεβαίως πρέπει να ασχοληθούμε με το κομμάτι των συναλλαγών του εμπορίου. Όμως δεν άκουσα από την Επιτροπή ότι μπορούμε να λύσουμε το θέμα της ιχνηλασιμότητας και της ε, σήμανσης ε, ετικετοθεσίας των προϊόντων που προέρχονται από την περιοχή αυτή της Δυτικής Σαχάρας. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες ε, καινούργιες λύσεις, αλλά ουσιαστικά είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση από τη στιγμή που δεν θέλει να αναγνωρίσει το Μαρόκο ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή περιοχή, ότι η Δυτική Σαχάρα δεν ανήκει στο Μαρόκο και εμείς πρέπει να αναγνωρίσουμε το θέμα της ε, κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτά τα καταχώμενα εδάφη. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες ε, προβάλλουν την αυτοδιάθεση μονίμως πλήττονται και διώκονται από τις ε, αρχές του Μαρακό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ τολμηρό να πούμε εδώ ότι έχει οριμάσει το θέμα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενσωματώσει σε αυτήν την συμφωνία και την ε, περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Θα κάνουμε λάθος αν πούμε κάτι τέτοιο. Και εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στα πλεονεκτήματα για τους πολίτες του Μαρόκο. Πρέπει να θυμάστε ποια ήταν η ουσία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και το έχει καθορίσει εξάλλου και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εδώ αναφερθήκαμε και στο ε, μέτωπο Πολυσάριο και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί οι επικοδομητικές λύσεις για αυτήν την ε, διαμάχη η οποία εδώ και δεκαετίες συνεχίζεται. Δεν μπορεί να έρθει από εμάς. Η δική μου ομάδα λοιπόν δεν θέλει να συμφωνήσει και να υπερψηφίσει. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν σίγουρα προσφυγές κατά της συμφωνίας αν αυτή εγκριθεί από εμά. Ναι. Θα είναι δύσκολο να φτάσουμε στη συμφωνία. Κυρία Μινέα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παραμένουμε στην ίδια κατάσταση. Είδαμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα. Έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορούμε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κόσμου εκεί, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Και το Πολυσάριο είναι ο επίσημος εκπρόσωπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι εδώ πέρα κάνει μια συζήτηση σημειολογίας. Λέει η Επιτροπή δεν έχει λέει ότι έχει σχέσεις με το Πολυσάριο, αλλά τελικά παίζει με τις λέξεις γιατί δεν έχει δώσει τη συγκαταθεσή του το Πολυσάριο. Είναι θέμα αξιοπιστίας όμως τελικά. Και επιπλέον υπάρχουν προϊόντα που φτάνουν στην Ευρώπη από αυτή την περιοχή και γι' αυτά δεν έχουμε καμία πρόταση. Τώρα λέτε ότι η νομική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά. Μα με κάθε σεβασμό σε αυτούς που εργάζονται στην ε, νομική υπηρεσία δεν είναι εκείνοι που αποφασίζουν. Εμείς αποφασίζουμε και πρέπει να τηρούμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το θέμα είναι το σχέσιο Πολυσάριο με Μαρόκο. Ο ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ, του κ. Γκουτιέρε, προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα. Ας αναβάλουμε την ψηφοφορία για αυτό το θέμα μέχρι να έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσει που γίνονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ τώρα που ξεκίνησαν και αυτό είναι το καινούργιο στην υπόθεση. Ευχαριστούμε. Η FDD. Ευχαριστώ την κυρία Λάλλοντ. Για το σχέδιο γνωμοδότησης, για την ε, Επιτροπή μας, νομίζω ότι πολύ σωστά περιγράφει το όλο θέμα των προβλημάτων με το Μαρόκο και την επέκταση στις εκτάσεις Δυτικής Σαχάρας. Νομίζω ότι σωστά επικεντρώνει οι συνάδελφοι, οι συνάδελφοι στις πτυχές της συμφωνίας που έχουν εμπορικό περιεχόμενο. Η συμφωνία δεν μπορεί να επιλύσει πολιτικά θέματα που πρέπει να λυθούν στο επίπεδο του ΟΗΕ. Υπάρχει όμως κατεπίγουσα ανάγκη να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με ένα τόσο σημαντικό σύμμαχο στη Μεσόγειο, στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και πολιτικής φύσης, για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Η πρόταση για εξομάλυνση και επειδή ε, από τους εκπροσώπους της Χάρας ξέρουμε ότι έχουν προωθηθεί γεωργικά προϊόντα προς την Ευρώπη και η ελληπής εφαρμογή της συμφωνίας με την περιοχή αυτή δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί δυσκολίες για τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι πρέπει να πάνε στο Αγκαντήρ σε πολλά χιλιόμετρα μακριά για την εξαγωγή των προϊόντων τους και αυτό αυξάνει πολύ το κόστος. Μάλιστα υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός από τους ίδιους ε, τους παραγωγούς του υπόλοιπου Μαρόκου. Η αποστολή που οργανώσαμε στο Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα είχε σκοπό ακριβώ να επιτρέψει προσωπικώ να λάβουμε γνώση του τι συμβαίνει σε αυτέ τι περιοχέ. Και μπορέσαμε να προσέξουμε ότι είναι πολύ ανεπτυγμένη η όλη περιοχή και από την πλευρά των υποδομών και των ε, ε, τεχνικών γνώσεων και τη γεωργική παραγωγή. Γι' αυτό η σύναψη συμφωνία με τη Δυτική Σαχάρα δεν μπορεί να είναι αρνητική για, για τον πληθυσμό της Δικής Σαχάρας ίσα ίσα θα ε, ωφελήσει και θα επιτρέψει την αναγνώριση των δικών μας γεωγραφικών αντίξεων στο Μαρόκο, ας πούμε. Ε, θα αποφύγουμε την παραποίηση και την πειρατεία. Και θα έχουμε διαφανέστερη εφαρμογή των συμφωνίων μα με το Μαρόκο για τον εντοπισμό των προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα. Θα προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε ένα σύστημα διακριτική μεταχείριση για του τοπικού παραγωγού και εργαζομένου. Και λίγα λόγια για τι διαφωνίε κάποιων συναδέλφων με ένα μήνυμα πριν από λίγε εβδομάδε. Πραγματικά λυπούμε που ε, στη συμμετοχή στην αποστολή στο Μαρόκο, δεν κατάλαβα γιατί υπήρχε πρόβλημα με την εκλογή τοπικών εκπροσώπων, ακόμα και με τη συμμετοχή υποψηφίων από το κίνημα Πολυσάριο. Αφιερώσαμε τρει ώρε συναντήσεων με 30 εκπροσώπους ε, τη κοινωνία των πολιτών ε, που ε, είναι εκπρόσωποι του Πολυσάριο, άλλους που είναι από το Μαρόκο και δεν ε, συμφωνούν με τη συμφωνία, διαφωνούν, αλλά πήγαμε και σε άλλες πόλεις Δυτικής Σαχάρας. Όλα αυτά έγιναν για να σεβαστούμε το στόχο της αποστολής μας και τους στόχους ε, της Επιτροπής Εμπορικών Θεμάτων. Ε, συναντήσαμε εκπροσώπους των παραγωγών, κυρίως εξαγωγέων, και ε, είδαμε και θέματα που μπορεί να άπτονται και των αρμοδίτων των άλλων επιτροπών. Α, αλλά δεν επικεντρώσαμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπούχνερ. Vielen Dank. <clears throat> Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω. Είπατε ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη. Εγώ νομίζω δεν είναι περίπλοκη η κατάσταση. Είναι ουσιαστικά μια χώρα, το Μαρόκο, η οποία κατέχει ένα συγκεκριμένο τμήμα το οποίο δεν ανήκει στη δική της επικράτρια και θέλει να υποφεληθεί από αυτό. Αν κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά τι λέει η έκθεση, όπως είπαν και άλλοι πριν από μένα, ουσιαστικά δεν είναι σκοπός της έκθεσης να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη, αν θέλετε, των πολιτών, του λαού που ζουν σε αυτή την περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αν διαβάσουμε προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου θα το διαπιστώσουμε ότι αναφέρεται. Και ένα δεύτερο σημείο που για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εάν δεν συνάψουμε αυτή τη συμφωνία, εμείς πλήττουμε τους πολίτες επιτόπου, γιατί ουσιαστικά εμποδίζουμε τις εξαγωγές. Δυστυχώς έτσι έχει η κατάσταση. Και αυτό που έμαθα πολύ πρόσφατα είναι ότι η, ο τοπικός πληθυσμός που ζει στη Δυτική Σαχάρα δεν είναι ένας ατόφιος πληθυσμός. Υπάρχουν έπικοι, υπάρχουν μαροκινοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί εκεί και υποφελούνται τελικά από αυτή την ανάπτυξη. Οι ντόπιοι ουσιαστικά έχουν απασχόληση τρίτης κατηγορίας ε, τους εκμεταλλεύονται οι Μαροκινοί, αυτοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί εκεί και εποφελούνται από την ε, ενδεχόμενη ανάπτυξη. Και πραγματικά, αν υπογράψουμε τη συμφωνία, δεν ξέρω ποιον θα πλήξουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, η Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λαλόντου για την ε, μέχρι τώρα εργασία που έχει Κοιτάξτε, συζητούμε για τη συμφωνία, αλλά η απόφαση του δικαστηρίου είναι σαφής. Είναι παράνομη η συμφωνία. Είναι ξεκάθαρο, γιατί πρέπει να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας. Δεν είναι λοιπόν νόμιμη η εισαγωγή, αν θέλετε, ε, προϊόντων από την περιοχή αυτή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Προσπαθούμε λοιπόν να συμμορφωθούμε με, το, με την απόφαση του δικαστηρίου. Και το πρώτο ερώτημα από το δικαστήριο είναι η σύμφωνη γνώμη ναι ή όχι των ντόπιων πληθυσμών και η δεύτερη είναι ότι ουσιαστικά δεν καλύπτει την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας αυτή η συμφωνία. Απλώς μπορεί να καλύψει τα προϊόντα. Πρώτον λοιπόν πρέπει να λύσουμε το θέμα της σύμφωνης γνώμης. Άκουσα τι είπε η Επιτροπή, ότι έγιναν διαβουλεύσεις. Η νομική υπηρεσία όμως η δική μας λέει ότι αυτό δεν αρκεί. Δεν ξέρουμε βεβαίως ξεκάθαρα βάσει της απόφασης του δικαστηρίου πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η σύμφωνη γνώμη των πολιτών. Από τη στιγμή λοιπόν που η απόφαση λέει ότι δεν καλύπτει τα προϊόντα της περιοχής της Δυτικής Σαχάρας εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Άρα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε την προέλευση των προϊόντων. Ξέρετε ότι η αρχή αυτή, το Μαρόκο δηλαδή, που ουσιαστικά ζητούμε αυτή τη στιγμή να μας δώσει στατιστικά στοιχεία, έχει την απόλυτη εξουσία σε αυτή την περιοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να βασιστούμε στις πληροφορίες που μας δίνει η αρχή του, ε, αυτή, το Μαρόκο δηλαδή. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και μηχανισμοί έτσι ώστε να ανατρέξουμε στην προέλευση των προϊόντων. Με κωδικούς παραδείγματο χάρη. Ένας μηχανισμός αξιόπιστος έτσι ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε στην προέλευση των προϊόντων για μία περιοχή η οποία δεν είναι αυτόνομη. Και αναφέρομαι στη Δυτική Σαχάρα. Δεν θέλω να κυρώσουμε μία συμφωνία χωρίς προηγουμένως να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και να βάλουμε σε ένα ψήφισμα κάτι αναθεώρηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι ρήτρε αναθεώρησης δεν έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πέσαμε στην παγίδα μια πρώτη φορά, δεν πρέπει να ξαναπέσουμε μια δεύτερη φορά, γιατί πραγματικά η αξιοπιστία μας σαν ε, μέλη του Κοινοβουλίου πλήττεται ανεπανόρθωτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να και εγώ ε, κ. Σούστερ, μπορώ να συμφωνήσω και εγώ θα ήθελα να ξέρω αυτός ο μηχανισμός για να ανατρέξουμε στην προέλευση είναι καθοριστικό σημείο. Δεν ξέρω αν μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου θα προλάβουμε να έχουμε αυτές τις απαντήσεις και όχι να βασιστούμε σε ό,τι μας λέει το Μαρόκο ή να πούμε θεωρητικά μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να μας βοηθήσει να δούμε την προέλευση των προϊόντων. Όχι άκουσε επίσης την ανάγκη ύπαρξης της σύμφωνης γνώμης της, του πληθυσμού επιτόπου. Δεν ξέρω, έχετε συζητήσει εσείς από την Επιτροπή και με εκπροσώπους του Πολυσάριου. Νομίζω η απάντηση είναι όχι. Και το επόμενο ερώτημά μου είναι, λέτε ότι είχατε επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων τι είπε συγκεκριμένα, ποια είναι η άποψή του. Εκείνος είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας ή κατά. Γιατί πραγματικά εν μέσω μιας διαμάχης την οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε, είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς, αν θέλετε, τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συμφωνίας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να μας πει εκείνος που ξέρει καλύτερα την κατάσταση. Τρίτον, γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ, μπορείτε να μου πείτε. Έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Μήπως πρέπει να περιμένουμε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο μέχρι τότε ίσως αυτή η διαπραγμάτευση έχει προχωρήσει. Και τότε θα αποφασίσουμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Αν ναι ή όχι πρέπει να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Δεν ξέρω, ε, νιώθω ότι αν θέλετε, αυτή τη στιγμή κάνουμε σαν μία εμπορική συμφωνία να μην είναι καθόλου πολιτική. Δεν είναι σωστό αυτό. Υπάρχουν ε, συγκρούσεις στην περιοχή, πολύ σοβαρά πολιτικά θέματα. Δεν είναι λοιπόν ουδέτερο το θέμα της εμπορικής συμφωνίας. Η Επιτροπή βεβαίως κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα καθαρά τεχνικά. Ναι, και η τεχνική όμως είναι πολιτική. Το ήθελες να μας πεις. Ο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για κάθε συμφωνία ισχύει αυτό, έτσι. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα και λίγες απαντήσεις. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Βεβαίως είμαστε συν Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ πρόκειται για θέματα που αφορούν ε, το δίκαιο, αλλά όχι μόνο το δίκαιο των επιχειρήσεων. Δεν είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Συμφωνώ απολύτως, είναι πολύ γενικότερο και φυσικά εδώ μπαίνουν και θέματα δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβάζω, πρέπει να διαπραγματευτεί με το Πολυσάριο για να μπορέσει να επιτύχει την ε, σύμφωνη γνώμη, τη συμφωνία των πολιτών της Δυτικής Σαχάρας. Δηλαδή θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει αυτή η σύμφωνη γνώμη για οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία η οποία θα πρέπει και θα μπορεί να εφαρμοστεί στην Δυτική Σαχάρα. Και αυτό θα καθορίσει αν ναι ή όχι θα τους πλήξει ή θα είναι χρήσιμο για αυτούς. Διαβάζω αυτή την παράθεση γιατί νομίζω ότι είναι καθοριστικό αυτό το σημείο. Είναι το, το κέριο ερώτημα, αν θέλετε, που προκύπτει διαβάζοντας αυτή την ε, έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία μας. Και βεβαίως ε, υπήρξε ε, επίσκεψη στην περιοχή, αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί τους οποίους κατονομάζει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σαν εκπροσώπους ζητήθηκε η γνώμη τους, ανεκφράστηκαν, θα είναι χρήσιμο για αυτούς, δεν θα είναι χρήσιμο για αυτούς. Αυτό είναι το άλλο συμπληρωματικό ερώτημα, καθοριστικό και αυτό. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί εδώ να παρακάμψει την πολιτική, αν θέλετε, τοποθέτηση γιατί είμαστε υπεύθυνοι για μία συμφωνία η οποία θα πρέπει με διαφάνεια και υπευθυνότητα να επεξεργαστεί, είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάμπαλικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επισημάνω ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν να δικαιώσει τους ανθρώπους της Δυτικής Σαχάρας. Και όμως, όμως εκπρόσωπος της Δυτικής Σαχάρας και ε, η εκπρόσωπη της κοινωνίας των πολιτών της Σαχάρας είναι αρνητική προς τη συμφωνία αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι ο μηχανισμό τεχνικό για την ε, καταγραφή των προϊόντων και τη προέλευσή του από την Δυτική Σαχάρα πρέπει να τελειοποιηθεί πριν εγκρίνει τη συμφωνία το Ευρωκοινοβούλιο. Η Δυτική Σαχάρα δεν είναι τμήμα του Μαρόκου. Θα πρέπει λοιπόν οι προσπάθειέ μα εντοπισμού των προϊόντων και τη προέλευσή του, αυτό ο μηχανισμό εχνηλασιμότητα, να γίνει ένα φόρουμ συνομιλίων και περαιτέρω πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω περισσότερα για τα επόμενα βήματα σε σχέση με την εχνηλασιμότητα όχι μόνο από την πλευρά του Μαρόκου, αλλά και από την πλευρά των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους. Πολλές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω η Σαμπίνε Χένσλερ να έχει σωστές και εύστοχες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια την κυρία Λαλόν για την ε, επιμελέστατη και πληρέστατη έκθεσή της για τόσο ευαίσθητο θέμα. Καλώς ορίζουμε την έκθεση που έχει συνταχθεί. Επίσης να θυμίσω την σημασία της συμφωνίας αυτής για την σταθερότητα της επενδύσεις στην περιοχή, για την συνεργασία τη συνεργασία πέραν των εμπορικών με, την, με τον πληθυσμό του Μαρόκου αλλά και της Δικής Σαχάρας, κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα και εξελίξεις. Ακούσαμε πολλές εκκλήσεις για την εχλασιμότητα. Και να βρει μια καινοφανή, μια ρηξικέλευτη λύση για τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τρεις διαφορετικές ε, ε, έννοιες που προέκυψαν από τη σημερινή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, η χνηλασιμότητα μέσω μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτός ο μηχανισμός προβλέπεται στη συμφωνία με το Μαρόκο την ίδια και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών τουλάχιστον ε, άπαξ μέσω της Επιτροπής Σύνδεσης. Αυτή τη στιγμή συζητούμε με το Μαρόκο του ομολόγου μας του Μαρόκου τι δυνατότητες να καθορίσουμε από τώρα το περιεχόμενο αυτών των ανταλλαγών. Συνολικά, αυτή τη στιγμή το Μαρόκο συμφωνεί με την πρότασή μα και η ανταλλαγή θα καλύπτει όλα τα θέματα που αναφέρει η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δίκτυα για την ανάπτυξη τη περιοχή, βιωσιμότητα, παραγωγή, εξαγωγέ των βασικών προϊόντων, φυτά προ καλλιέργεια και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λεπτομερέστατες πληροφορίες σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να λειτουργήσει το αργότερο δύο μήνες μετά τη θέση ισχύ τη συμφωνίας. Περιμένουμε όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και νωρίτερα και να ξεπεράσουμε τα προγνωστικά. Δεύτερο σημείο, δεύτερη έννοια και νομίζω ότι αυτό απαντά περισσότερο τις ερωτήσεις της κυρίας Αρενά και άλλων. Αυτή τη στιγμή συζητούμε με το Μαρόκο έναν μηχανισμό τεχνικού χαρακτήρα για να μπορέσουν τα στοιχεία για τις εξαγωγές να καταγράφονται αυτομάτως και να συλλέγονται πληροφορίες για τις εξαγωγές, τα προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα. Αυτό θα μας επέτρεπε να καταγράψουμε στατιστικά σε πραγματικό χρόνο το τι συμβαίνει. Όχι αναδρομικά, ούτε κατόπιν εορτής. Ή όπως συμβαίνει με τον μηχανισμό που περιέγραψα προηγουμένως το θέμα το μελετούμε σε τεχνικό επίπεδο και ελπίζουμε ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορεί να λειτουργήσει πολύ γρήγορα. Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με το Μαρόκο για το συγκεκριμένο σημείο και είμαι βεβαία ότι λύση θα βρεθεί και μάλιστα γρήγορα. Τρίτον, η επισήμανση των προϊόντων. Το είπατε πολλές φορές. Να είμαι σαφής. Το θέμα της επισήμανσης είναι εκτός του πεδίου αυτής της εμπορικής συμφωνίας. Είναι σαφές ότι οι εισαγωγέ προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, πληρούν τους όρους και τις προθέσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όμως η ετικετοθεσία είναι εκτός της συμφωνίας. Αυτό που κοιτάζουμε είναι ο πρώτος μηχανισμός που ανέφερα ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο άθρησης των πληροφοριών, συνόλων πληροφοριών, όχι μία-μία, και μετά ένας μηχανισμός σε πραγματικό χρόνο ε, ταυτόχρονης καταγραφής της προέλευσης και των ε, εισαγωγών. Προχωρούμε ως το δυνατόν πιο γρήγορα σε συνεργασία με τους μαροκινούς εταίρους, οπότε το Κοινοβούλιο θα έχει μια συνολική τελική εικόνα για τη συμφωνία και τη μορφή θα πάρει όταν θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι ζωτική σημασία στοιχείο για το Κοινοβούλιο. Συνάντηση με τους Μαροκινούς διαπραγματευτές έχουμε μεθαύριο ήδη και ελπίζω εκεί να προκύψουν καλές ειδήσει για να σας τις μεταφέρουμε σύντομα. Επίσης, να αναφερθώ σε μερικά από τα άλλα σημεία που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτα απ' όλα το θέμα της σύμφωνης γνώμης. και άνα διαδικασία της σύμφωνης γνώμης καλύπτει τις απαιτήσεις του δικαστηρίου. Να σας παραπέμψω στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό που λέει ότι η διαδικασία των διαβουλεύσεων απηχεί ε, βήματα που θα μπορούσαν ε, ε, εύλογα να θεωρηθούν ως προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών τη Δυτική Σαχάρα. Το δικαστήριο λοιπόν δεν μα είπε πώ πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά όπω είπε και η νομική σα υπηρεσία, κάναμε ό,τι είναι λογικό δυνατό και εφικτό για να πετύχουμε να έχουμε σύμφωνη γνώμη. Σε ό,τι αφορά το τι εκπροσώπηση έχει ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας στο μέτωπο Πολυσάριο, θα σας παραπέμψω στην ομοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, σημείο 24, όπου λέγεται ρητός από την νομική υπηρεσία και ορθώς, ότι το ψήφισμα του ΕΕ δεν ασχολείται με τον ορισμό των ανθρώπων, ούτε με, την, με το δικαίωμα και την νομιμοποίηση να εκπροσωπεί κανεί το λαό. Γιατί τώρα το μέτωπο Πολυσάριο στις πολιτικές διαδικασίες θεωρείται ως ε, εκπρόσωπος είναι γιατί δεν υπάρχει σαφής ορισμός του λαού, των ανθρώπων που εκπροσωπεί το Πολυσάριο. Και εν τέλει, γιατί δεν κάνουμε το ένα και το άλλο με το Πολυσάριο, σε άλλα κομμάτια της επικράτειας. Αυτό που χρειαζόμαστε και μάλιστα χρειάζεται και το συγκεκριμένο κοινοβούλιο είναι να έχουμε μια αξιόπιστη τελωνιακή αρχή για να μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι οι προτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται σεβαστές. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα ελέγχου των τελωνιακών αρχών. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε προβλήματα με τους ιδίους πόρους και με την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και ότι δίνουμε προτιμήσεις εκεί που δεν πρέπει. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό από την τελωνιακή σκοπιά να έχουμε αξιόπιστες αρχές. για την περιοχή για την οποία παρέχουμε προτιμήσεις. Ευχαριστώ. Έχω τρεις επερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι και επί του θέματος. Κυρία Χάουταλα. Όταν λέει η Επιτροπή ότι το θέμα της σήμανσης είναι εκτός πεδίου εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, θέλω να τονίσω ότι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εντοπίζουν τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Πώς μπορείτε να εγγυηθείτε λοιπόν ότι τηρούνται και προστατεύονται τα δικαιώματα αυτά των καταναλωτών. Άμα επιταδούμε το διεθνές δίκαιο, νομίζω ότι ελάχιστοι εδώ μέσα θα λέγανε ότι είναι φυσιολογικό να έχει κανείς εμπορική συμφωνία με τη Ρωσία ε, ή την Κρυμαία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό ζήτημα διεθνούς δικαίου και δεν λαμβάνεται αρκετά σοβαρά υπόψη. Έχω την εντύπωση ότι και η Επιτροπή αλλά και οι περισσότερες πολιτικές ομάδες, ακόμα και διχασμένες κάποιες από αυτές μεταξύ τους, τελικά θέλουν να τα έχουν όλα και την μπίτ ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θέλουμε τους όλους. Ναι, και εγώ Έχω μια ερώτηση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει στη δικιά της λογική. Μα ακριβώς αυτό είναι που συζητάμε. Δεν έχετε απαντήσει. Γιατί επιμένετε να ακολουθείτε αυτό το δρόμο. Γιατί δεν είσαστε σε θέση να κάνετε διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα ζητήματα και να βρείτε μία λύση υπέρ των ενδιαφερόμενων μερών. Εσείς εξακολουθείτε με όλα τα σενάρια που περιγράφετε, παραμένετε στην ίδια λογική η οποία είναι στραβή. Γιατί επιμένετε. Ευχαριστώ. Θέλω να πω και εγώ ότι κατάλαβα καλά ότι το μέτωπο Πολυσάριο είναι κατά Εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε από τη δικιά μας την πλευρά. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι το μέτωπο Πολυσάριο είναι η νόμιμοι εκπρόσωποι της Δυτικής Σαχάρας. Γιατί. Μπορείς να μας το πει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Ηνωμένα Έθνη διαπιστώνουν ότι η ομάδα επίσημα αναγνωρισμένη λέει όχι. Ε, ποια είναι η συνέπεια αυτού του γεγονότος για μας και για την Κομισιόν. Αυτό ήθελα να πω και πριν. Ο ειδικό αποσταλμένος στο ΙΕ τι έχει να πει γι' αυτό. Θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα να ολοκληρωθεί η συμφωνία ή λέει όχι θα επιδεινωθεί η κατάσταση ή θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή θα μπορούσε αντίθετα να βοηθήσει να σταματήσει η διένεξη. Εδώ ακούμε διπλωματικό λόγο, ρητορική, δεν είναι αυτά που χρειαζόμαστε εδώ. Ωραία. Ίσως να ακούσουμε την απάντηση. Okay. Uh, let me just uh, in reply to Mrs. Hotala. Ευχαριστώ προς την κυρία Χαουτάλα για τη σήμανση. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία και ισχύει για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Και το ίδιο θα ισχύσει και για τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας. Δεν θα υπάρξει διαφορετική ρύθμιση από αυτού. Για το πολυσάριο. Τώρα το μέτωπο πολυσάριο. Επιτρέψτε στο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά προηγουμένως από την Ταξούντ ο συνάδελφος θέλει να προσθέσει κάτι ως απάντηση. Ναι, ευχαριστώ. Γιατί ακολουθούμε αυτή τη λογική που ρώτησε ο κύριος Σόλτς. Μα ένα μόνο τρόπο έχουμε βρει να προσφέρουμε προτιμήσεις στις εισαγωγές από τη Δυτική Σαχάρα. Δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική. Δεν έχουμε υπόψη μας κάποια άλλη δυνατότητα κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες. Ωραία, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τώρα. Οι διαβουλεύσεις συμπεριέλαβαν και το Πολυσάριο, τουλάχιστον από τη δικιά μας ε, την πλευρά αυτό θέλαμε. Εξάλλου, διάφοροι άλλοι μη κυβερνητικοί εταίροι συμμετείχαν, όπως και εκλεγμένες αρχές του Μαρόκου και το Περιφερειακό Συμβούλιο και αντίστοιχες αρχές της Δυτικής Σαχάρας. Οπότε, εμείς προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με το Πολυσάριο για αυτό το ζήτημα, για το κατά πόσο θα δώσουν τη σύμφωνη γνώμη όχι. Δεν ανταποκρίθηκαν όμως θετικά στην πρόσκλησή μας που έγινε επανειλημμένος. Δεν είχαμε ούτε απάντηση, ούτε αποδοχή της πρόσκλησης. Αυτή λοιπόν είναι η απλή απάντηση στην ερώτηση. Το Πολυσάριο μετά την πρώτη φορά προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί τους, εξέδωσαν ένα κοινοθέν τύπου όπου ξεκαθαρίζουν ότι δεν συμφωνούν με αυτή τη συμφωνία, όχι εξαιτία τη συμφωνία αυτή καθεαυτή του περιεχομένου, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του θεωρεί τον μόνο συνομιλητή για τι διαπραγματεύσει αυτές. Δεν αρνούνται δηλαδή την ουσία, την χρησιμότητα της συμφωνίας, αλλά για λόγους πιο πολιτικούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρήσει ότι ο μόνος συνομιλητή της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι το πολυσάριο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ο λόγο είναι απλός και είναι ότι καμία χώρα μέλος, εκτός ίσως από κάποιες εξαιρέσεις, και οι περισσότερες χώρες του ΟΗΕ δεν αναγνωρίζουν το Πολυσάριο, ούτε την δημοκρατία που έχει ανακηρύξει την Αραβική Δημοκρατία το Σαροή δεν το αναγνωρίζουν. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν προβαίνουμε σε διαπραγματεύσεις αυτού του τύπου. Η πολιτική πραγματικότητα με τη διπλωματική προτεραιότητα βασίστε σε αντικειμενικά στοιχεία. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σχολιάσω και σε δύο πράγματα που είπαν οι ευρωβουλευτές. Πρώτον, τι σκέφτεται ο ΙΕ για όλα αυτά και γιατί να βιαστούμε για αυτή την ψηφοφορία. Για το πρώτο. Κάποιοι από εσά θα ακούσατε τον κύριο Χορσκούλερ να ε, μιλάει και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην ΙΝΤΑ πριν από λίγους μήνες. Και ο ΙΕ δεν πήρε θέση. Η μόνη τοποθέτηση ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πλευρές θα έπρεπε να σέβονται το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τους νόμους και θα έπρεπε να δρουν με τέτοιο τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την διαδικασία του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα. Η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι τώρα ανταποκρίνεται απόλυτα σε αυτές τις προϋποθέσεις που βάζει ο ΙΕ. Δεν ε, ζημιώνει, δεν είναι ασύμβατη με την νομοθεσία του ΙΕ. Γιατί να βιαστούμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία και δεν περιμένουμε την 4η Δεκεμβρίου, ρωτάτε. Μα μην ξεχνάμε ότι οι συζητήσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 4 και 5 Δεκεμβρίου στη Γενέβη, αυτές θα είναι οι πρώτες σε μία δεκαετία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να είναι οι τελευταίες συναντήσεις αυτές. Πρόκειται για μία μακρά διαδικασία μεταξύ ε, μερών, των οποίων οι θέσεις είναι αντιδιαμετρικά αντίθετες και θα πάρει ναι. χρόνο να μειωθούν αυτές οι διαφορές μεταξύ τους και να επιτευχθεί κάποια συνένεση για μια αποδεκτή από τις δύο πλευρές συμφωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συνάντηση της 4ης Δεκεμβρίου αποτελεί ένα μόνο βήμα. Αν να βάλετε τη δικιά σας απόφαση μέχρι τότε δεν θα έχετε καμιά ξεκάθαρη εικόνα. Θα πρέπει να περιμένετε μάλλον την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχει ξεκαθαρίσει κάπως η εικόνα. Καλώ ευχαριστούμε η συγκήτρια κυρία Λαλόντ. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω πρώτα απ' όλα στη διαδικασία του ΟΗΕ. Υπήρξε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 2285 νομίζω πριν από δύο μέρες για την παράτηση της Μινουρσό της αποστολής για έξι μήνες αντί για ένα χρόνο. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα επιταχύνεται γιατί θα πρέπει να έχει βρεθεί μια λύση πριν την 30η Απριλίου. Αυτό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που περιπλέκει ε, το θέμα. Έπειτα, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους εκπροσώπους του κ. Κολέρ και θα υπάρξει και νέα συνάντηση. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος. Δεν μας είπαν ποτέ ότι πρέπει να περιμένουμε ε, την 4η 5η Δεκεμβρίου για να προχωρήσουμε τις δικές μας διαδικασίες και να ψηφίσουμε στην ίντα. Γιατί πρόκειται για δύο χωριστά πράγματα. Ήταν ξεκάθαρη σχετικά με αυτό. Και από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Κολέρ, και οι ίδιοι κάνανε μία αποστολή επιτόπου και έχω την αίσθηση ότι αποκόμισαν την ίδια αίσθηση όπως και εμείς όσον αφορά τις οικονομικές προϋποθέσεις, περιβαλλοντικές, από τις οποίες εποφελείται ο κόσμος της Δυτικής Σαχάρας, γιατί πρόκειται για τόπους. Δεν νομίζω ότι τους φέρανε από το Μαρόκο, είναι Σαχαροή. Το λέω και στην έκθεσή μου πολλές φορές. Μας εκπλήσει η οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή να την παραβλέψουμε. Για να πατήσω τώρα και στη Μαρία Αρενά. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στο θέμα της συχνηλεσιμότητας, γιατί είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια προϊόντα προέρχονται πράγματι από τη Δυτική Σαχάρα φαντάζομαι θα τσακωθούμε σε αυτό με τους Μαροκινούς γιατί δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι συμφωνούν. πιστεύουμε όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα πρέπει να πετύχει από το Μαρόκο να δεχτεί τη σωστή διαδικασία αναγνώρισης των προϊόντων. Πρέπει να ξέρουμε ποια προϊόντα προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και ποια όχι. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι τα πάμε όλα. Ελπίζω να πάτησα σε όλους και στην κυρία Χαουτάλα να πω κάτι. Ειλικρινά στην διερευνητική μας αυτή αποστολή, όπου ήμασταν τρεις από το EFTT, η κυρία Μπεγκίν, η κυρία Χαουτάλα και εγώ ίδια, δεν μας δόθηκε εντύπωση κατά τη διάρκεια της αποστολής, τουλάχιστον για την κυρία Μπεγκίν και για μένα σίγουρα μπορώ να μιλήσω, ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε χαροή από τις επαφές Πολυσάριο ε, μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Να ξέρετε ότι πέρασαμε πάρα πολύ ώρα και με του μεν και του δύο. Η κυρία Χωτάλ έφυγε με στη νύχτα για να συναντήσει άλλους φορείς. Φαντάζομαι ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ε, βγάλαμε κανένα συμπέρασμα. Δεν ξέρω βέβαια τι συνέβη με εκείνη εκεί που πήγε το ξημέρωμα. Αυτή είναι η ανάλυση μου. Μια τέτοια οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τη διαδικασία του κ. Κολέρ. Θα δούμε τι θα γίνει και στη Γενέβη και θα πάνε γρήγορα τα πράγματα γιατί 30 Απριλίου, αν δεν υπάρξει νέα παράταση της αποστολής, οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να τελειώσουν με αυτή την υπόθεση που κρατάει τόσο καιρό. Θα βρεθεί μια λύση. Οι Μαροκινοί επίση θα αναγκαστούν να κάνουν μια προσπάθεια για το θέμα της συχνηλασιμότητα. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία η οποία να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Η κυρία Χαουτάλα θέλει να εξηγήσει τι έκανε μέσα τη νύχτα, τη βαθιά νύχτα, το ξημέρωμα επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου και θέλω και δικιά μου εμπειρία να αναφερθεί στην έκθεση, αλλά μου είπαν ότι επρόκειτο για μια ε, προσωπική ιδιωτική παρατήρηση και δεν έχει καμία σχέση με την ε, αποστολή μας. Όμως μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι οι οργανώσεις των πολιτών που βρίσκονται υπέρ της αυτοδιάθεσης είναι θύματα όχλησης. Όντως, μεσάνυχτα με δύο τα ξημερώματα υπήρχαν πάρα πολλοί αστυνομικοί, σταμάτησαν το αυτοκίνητο, το κατηγόρησαν τον οδηγό ότι δεν φορούσε ζώνη και του αφαίρεσαν την ε, αδειοδήγηση. Συζητήσαμε με τους αστυνομικούς την παρουσία πολλών αυτοκινήτων της ε, αστυνομίας αλλά, πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι η έκθεση που με κάθε σεβασμό συνέταξε η κυρία ε, Λαλόντ είναι μονόπλευρη και δεν περιλαμβάνει τίποτα, καμία παρατήρηση που θα μπορούσε να προσταθεί για τα όσα είδαμε και συναντήσαμε στο Γιάννου και στην Τάκλα. Πρόεδρος, είναι διαφορετικές απόψεις. Προθεσμία. 7 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι για υποβολή τροπολογιών. 7 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ωραία. Και έτσι ολοκληρώθηκε η... τα σημεία αυτά. 18. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Μια σύντομη παρατήρηση του κυρίου Προύστ για το συνεχιζόμενο τριμερή διάλογο. Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να πω για τη μέθοδο ε, παρακολούθησης των επενδύσεων Έχουμε παραμείνει στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά θέλω να εξηγήσω σε ορισμένου συναδέλφου ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τι προτεραιότητέ μα ω Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε πετύχει συμφωνία για τα κλάστερ 1 και 2, κλάστερ όπου κυρίω ε, θα ε, καθοριστεί η αρχιτεκτονική των μελλοντικών μας συστημάτων και τη συνεργασία στα θέματα των ξένων επενδύσεων. Τριμερή διάλογο έχουμε οργανώσει και για αύριο που θα αφορά το τρίτο κλάστερ και θα δούμε τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι τεχνολογίε για τι υποδομές, τις στρατηγικές υποδομές και τα προγράμματα που θεωρούμε στατικής σημασία. και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση ότι είναι πολύ εποφελή, πολύ μάλλον καρποφόρηση οι δημοτεύσεις μα και ελπίζουμε θα οδηγηθούν σε αίσιο πέρα. Ξέρετε βέβαια ότι υπάρχουν κάποια θέματα που παραμένουν εκκρεμή και τα οποία είναι σημαντικά και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Και η δική μου αίσθηση είναι ότι οι διαπραγματεύσει μπορούν να πάνε καλά και πιστεύω ότι σωστά ε, έχω τέτοια αισιοδοξία. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εργάζεται αποτελεσματικά για να βρει συμβαστικέ λύσει και την Αυστρική Προεδρία με την οποία συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και στενά για να καταλήξουμε σε συμφωνία στο δυνατόν πιο γρήγορα. Διότι για τη συμφωνία αυτή το χρονοδιάγραμμα μου φαίνεται καθοριστική σημασία. Ε, de Okay, no questions to Mr. Proust. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Προύστ, οπότε περνάμε στο σημείο 20, διάφορα, τίποτα, επόμενη συνεδρίαση 19 και 20 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.